Θα ξεκινήσουμε, παρακαλώ καθίστε. Ε, καλησπέρα σε όλους σας. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε παρατηρήσει ή ενστάσεις για την ημερήσια διάταξη. Θεωρείται εγκεκριμένη λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Δεν έχω να σας κάνω κέρδιες ανακοινώσεις, απλώς θέλω να σας υπενθυμίσω ότι για τη σημερινή μας συνεδρίαση έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό γλωσσών προς τις οποίες διερμηνεύονται τα λεγόμενά μας. Περνάω στο επόμενο σημείο τώρα. Η Κομισιόν θα ήθελε να κάνει κάποια ανακοίνωση, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, η Κομισιόν δεν έχει να σας κάνει καμία ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μια ερώτηση του κυρίου Κόρτες Λάστρα προς την Κομισιόν για τη σημερινή μα συνεδρία. Βεβαίω, καφέ θέλω. Είναι η ερώτηση του κυρίου Κορτές Λάστρα που βρίσκεται στο φάκελό σας προσκαλώ την Κομισιόν να δώσει απάντηση. Ο κύριος Λιτβίν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απαντών στο ερώτημα του εντύμου αυτού μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορώ να σας πω ότι οι υπηρεσίες της Κομισιόν θέλουν να εκφράσουν την ικανοποίησή τους σε σχέση με την θετική ε, αξιολόγηση που εδόθη στο Eurosocial 2 από τις εξωτερικές υπηρεσίες αξιολόγησης. Είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό το 2007-2013 με συνολική χρηματοδότηση 40 εκατομμυρίων και θα ε, περατωθεί καταρχήν μέχρι το τέλος του 2015. Δεδομένου του ότι εξακολουθεί ο σχεδιασμός για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο είναι κάπως πρόωρο να σας δώσω λεπτομέρειες για τα σχέδια τα οποία θα μπορούσαν να τύχουν υποστήριξης <clears throat> για τα επόμενα χρόνια. Ακόμα δεν έχουν καθοριστεί κύριοι άξονε συγκέντρωση της χρηματοδότηση και συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με τι κυβερνήσει, με την κοινωνία των πολιτών, με το Ευρωκοινοβούλιο. Ε, έχουμε πάρει πολύ σημαντικά διδάγματα για τις μελλοντικές δράσεις μας από τα προηγούμενα προγράμματα του Aerosocial και φυσικά θα λάβουμε όλα αυτά υπόψη για τον προγραμματισμό στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πιστεύω θα πρέπει να εστιάσουμε σε ένα πιο περιορισμένο αριθμό τομέων, αλλά επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την κοινωνική συνοχή και τη μείωση των ανισοτήτων στη Λατινική Αμερική. Μέχρι το τέλος του 2015 λοιπόν θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα και πιστεύω ότι του χρόνου θα μπορούμε να έχουμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες όπως πολύ σωστά το επισημαίνει το έντιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κόρτες Λάστρα θέλετε να πείτε κάτι. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε όταν έκανα αυτή την ε, ερώτηση, όπου εξήρα και το το έργο του Εροσοσιαλ. Θα ήθελα να ακούσω από την Κομισιόν κυρίως το ότι θα διατηρηθεί συνέχεια σε αυτά τα προγράμματα και δεν θα σταματήσει η εφαρμογή του. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε τότε στο σημείο 5. Ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Τζόρτζεβα που θα έρθει ο Σονούπο. Έρχεται.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 Σε δύο λεπτά θα δει η κυρία Τζόρτζεβα, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Λοιπόν, έχει έρθει η κυρία Επίτροπο. Κυρία Επίτροπε, έχουμε μια αντάλλαγη απόψεων σε σχέση με τα ηλυμένα μέτρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μετά από τον τυφώνα που έπληξε τι Φιλιππίνες και χαιρόμαστε που μπορούμε να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων παρουσία της κυρίας ε, Τη της Επιτρόπου για την, ε, τα ανθρωπιστικά θέματα και την αντιμετώπιση των κρίσεων και επίσης είναι παρόν ο Γενικός ε, Διευθυντής της ε, Αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, ο κύριος Φρουκτουόζου Ντουμέλου. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις σας ενώπιον της Επιτροπής ανάπτυξης και ο λόγος για τον οποίο γίνεται σήμερα αυτή η ανταλλαγή απόψεων είναι ακριβώς να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του τυφώνα ο οποίος έπληξε τις Φιλιππίνες την προηγούμενη εβδομάδα. δεν ξέρουμε ακόμα πόσο μεγάλες είναι οι ανθρώπινες και ηλικίε ζημίες αλλά οι εκτιμήσεις τις αναφέρουν σε 5.535 νεκρούς, 20.000 ε, τραυματίες και πάνω από 100.000 αγνώμους. Και επίσης πάνω από ένα εκατομμύριο κατοικίες έχουν εν μέρη ή πλήρως καταστραφεί. Αλλά θα δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία Τσόζεβα, η οποία αμεσως στην κυρια τζοζεβα η οποια πηγε στις Φιλιππίνες μετά από την καταστροφή αυτή και ο κύριος Φουτουόσο Ντεμέλο θα λάβει το λόγο μετά την κυρία Επίτροπο και θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις και να λάβουμε απαντήσεις. Κυρία Επίτροπο, έχετε το λόγο. Euh, euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από μια πολύ μεγάλων διαστάσεων καταστροφή που έπληξε τις Φιλιππίνες. Ο χάρτης που βλέπετε ε, εδώ επάνω δείχνει τη διαδρομή ενός τυφώνα επίπεδου 5 τεραστίων, τεραστίας ισχύος που έπληξε μεγάλο τμήμα των Φιλιππίνων με ανέμους που έφτασαν σε ταχύτητα 325 χιλιόμετρα την ώρα. Οι Φιλιππίνες ε, κατασκεύασαν καταφύγιο για να προστατευθούν σε κέντρα εκένωσης ε, ε, οι άνθρωποι με βάση την υπόθεση ότι θα, έχει, θα είχε 160 χιλιόμετρα ταχύτητα την ώρα ο, ο άνεμος και ήταν στην πραγματικότητα διπλάσια η ταχύτητά του. Το πρόβλημα της αντίδρασης ε, είναι ορατό στο χάρτη. Η διάμετρος ήταν 50 χιλιόμετρα, πέρασε από μεγάλο αριθμό νησιών που κάποια είναι τα φτωχότερα νησιά των Φιλιππίνων. Όταν έφτασα πέταξα από πάνω από την περιοχή αυτή με μικρό ελικόπτερο και είδα εγώ η ίδια τη διαφορά μεταξύ των περιοχών των οποίων εφίσθη ο τυφώνας και των άλλων. Και η διαφορά είναι σαν να λέμε ανάμεσα στον παράδεισο και την κόλαση. Σειρά χωριών, μεγάλη, μεγάλος αριθμός χωριών καταστράφηκε ολοσχερός και η περιοχή που επλήγει περισσότερο είναι το Τακλομπάν, που είναι μια πόλη που γονάτισε. Εγώ την επισκέφθηκα μία εβδομάδα μετά τον τυφώνα. Και ακόμα στο δρόμο από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο της πόλης και από τις δύο πλευρές του δρόμου υπήρχαν μαύρες σακούλες που περιείχαν ε, νεκρούς και Ακόμη ε, πολλά θύματα δεν μπόρεσαν να ε, βρεθούν στα χαλάσματα. Σε αυτή την περίπτωση ε, είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδρασε ταχύτατα και σύντονα και αυτό που βλέπετε τώρα εδώ στο χάρτη είναι η επόμενη μέρα. Χτύπησε Παρασκευή ο τυφώνας. Το Σάββατο οι πρώτες διεθνείς ομάδες ε, αξιολόγησης είχαν φτάσει από την Ευρώπη και η Ανθρωπιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έστειλε αμέσως δύο ομάδες. Τη μία στην, στο, στο νησί ε, Λάιτι που επλήγει πιο πολύ από όλα τα άλλα και στο Μπόχολ. Νησί και αυτό. Γιατί, γιατί το Μπόχολ είχε πληγεί και από σεισμό μόλις δέκα μέρες πριν από την έλευση του τυφώνα και ανησυχούσαμε πολύ διότι εκείνοι οι άνθρωποι που είχαν τόσο σκληρά πληγή μία φορά ε, θα ε, πλήττοντο κι άλλοι. Ε, αυτό ευτυχώς δεν επαληθεύτηκε. Την επόμενη μέρα πήραμε την απόφαση να δώσουμε 3 εκατομμύρια ευρώ και αυτή ήταν η πρώτη οικονομική συμβολή ε, προς τα θύματα του τυφώνα ενώ οι εταίροι μας ήδη ε, προχωρούσαν στην παροχή της βοήθειας. Το, το Telecom Team από το Telecom San Frontier, Telecom χωρίς σύνορα, οι ομάδες τους έφτασαν στο Λάιτε την Πέμπτη, δηλαδή την ημέρα πριν ε, να χτυπήσει ο τυφώνας. Γιατί ξέραμε ότι θα ε, πλήττονται και οι τηλεπικοινωνίες ε, διότι το πλήγμα ήταν μεγάλης κλίμακας και έτσι δεν θα μπορούσαμε να παράσχουμε βοήθεια. Η ομάδα λοιπόν κατέστη επιχειρησιακή αμέσως μετά το χτύπημα του τυφώνα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την ανθρωπιστική παροχή βοήθειας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Την επόμενη μέρα αποστήλαμε ε, ομάδες αξιολόγησης στις πληγήσεις περιοχές μαζί με τα κράτη-μέλη, πάλι με απόλυτα συντονισμένο τρόπο και περηφανεύομαι για την Ευρώπη όταν πω ότι εμείς καλύψαμε χωρίς διακρίσεις όλη την περιοχή. Δεν στείλαμε δηλαδή ομάδες μόνο εκεί που ήταν οι δημοσιογραφικές κάμερες αλλά στείλαμε ομάδες ε, σε κάθε περιοχή όπου η ζημιά ήταν σημαντική. Και με βάση τη δουλειά μας που υποστηρίξαμε μάλιστα και την ομάδα των Ηνωμένων Εθνών και μπορέσαμε γρήγορα να ε, δούμε ποιες ήταν οι ανάγκες και να φροντίσουμε ότι η βοήθεια, δηλαδή ε, παροχή σε είδος και οικονομική βοήθεια, θα παράσχονταν με τρόπο συντονισμένο, ούτως ώστε να μην βοηθηθούν κάποιοι δυο φορές ενώ άλλοι καθόλου και βλέπετε στο χάρτη τις ανάγκες όπως κωδικοποιήθηκαν Και επίσης, όπως ακούσαμε από την κυρία Στρίφλερ, κατεγράφει τι ακριβώς συνέβη σε σχέση με απώλειες ε, ζωής, ε, ζημιές στον πληθυσμό, καταστροφή κατοικιών. Κινητοποίησαμε από την Ευρώπη μαζί με τα κράτη-μέλη ε, ένα γενναιόδωρο ποσό πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια, εκ των οποίων η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα βρίσκεται στα 23 εκατομμύρια ευρώ. 10 εκατομμύρια ανθρωπιστική βοήθεια, 10 εκατομμύρια ε, δόθηκαν από τον Επίτροπο Πίμπαλξ που ήταν την εποχή του τυφώνα για ταχεία αποκατάσταση και 3 εκατομμύρια για συγχρηματοδότηση ε, από τα κράτη-μέλη. Μπορέσαμε να βοηθήσουμε άμεσα καλύπτοντας τις ε, άμεσες ανάγκες. Έγινε ε, βοήθεια διανομής τροφίμων, ε, διανομή και καθαρισμός, διανομή ε, καθαρού ύδατος, ε, ιατροφαρμακευτική βοήθεια και καταφύγια, στέγη, καταβλισμοί. βέβαια εδώ έχουμε ένα πίνακα δυσανάγνωστο, αλλά πολύ χρήσιμο, γιατί για πρώτη φορά σε μια τέτοια μεγάλη έκτακτη ανάγκη Είχαμε εξαιρετική συνεργασία και συντονισμό με τα κράτη-μέλη μας και σαφή συμβολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για υποστήριξη των προσπαθειών σε τοπικό επίπεδο και σε, υποστηρίζοντας και τα Ηνωμένα Έθνη. 22 κράτη-μέλη συνέβαλαν στη συνολική αυτή προσπάθεια κάποιοι ε, μόνο με οικονομική βοήθεια, ε, άλλοι σε είδος, άλλοι και τα δύο. Πάντως η Ευρώπη έδρασε συνολικά και το σύνολο ε, έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα παραπάνω από το άθροισμα των μερών. Κάποια συμπεράσματα τώρα με βάση αυτά που κάναμε μέχρι τώρα και δύο λόγια σχετικά με τα επόμενα βήματα. Πρώτον, για άλλη μια φορά ξεκάθαρα βλέπουμε ότι αυτό που ήταν ένα τυχαίο και σπάνιο γεγονός μιας πολύ μεγάλης καταστροφής τώρα γίνεται σχεδόν ένα γεγονός σε αιτήσια βάση. Τα τελευταία χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο είχαμε μία καταστροφή ε, μεγάλη φυσική καταστροφή, καμιά φορά και δύο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχτούμε ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στην ετοιμότητα και την πρόληψη, γιατί ο κόσμος μας ζητάει περισσότερα από μας πλέον. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι συνεργαστήκαμε με τις Φιλιππίνες ως μια χώρα που ε, έχει πολλές, τάση για πολλές καταστροφές στον τομέα της ετοιμότητας 7 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας το, ε, το επενδύσαμε για πρόληψη ε, και εκεί και σε άλλες ευάλωτες περιοχές. Δεύτερον, Βλέπουμε πόσο ωφελεί το καινούριο κέντρο μας συντονισμού της ε, ε, κατεπίγουσας βοήθειας. Αν δεν το έχετε επισκεφθεί, σας συνιστώ να το επισκεφθείτε γιατί είναι η καρδιά του συντονισμού. Έτσι μπορούμε να συνδυάζουμε δορυφορικά δεδομένα με τις δυνατότητες του κοινού κέντρου έρευνας για να προβλέψουμε τι θα συμβεί και μετά να κινητοποιήσουμε την αντίδρασή μας με τρόπο μαζικό και καλά συντονισμένο. Ο συντονισμός και η συνεργασία στην Ευρώπη ιδιαίτερα σε εποχή όπου είναι περιορισμένοι πόροι και μεγάλες είναι ανάγκες, είναι απόλυτα αναγκαία, αναγκαίος. Και απευθύνομαι εδώ στο Κοινοβούλιο που μας ζήτησε να κάνουμε περισσότερα πράγματα σε αυτό το τομέα. Σε μια εβδομάδα από τώρα, σε 8 μέρες από τώρα, το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει τη νέα νομοθεσία για την πολιτική προστασία η οποία νομοθεσία θα βάλει επίσης όρους την ε, δράση και την πρόληψη και την ετοιμότητα. Τώρα, για να ξαναγυρίσω στις Φιλιππίνες, ακόμα είμαστε στη φάση της παροχής ε, ε, μέτρων ανακούφισης. Συνεχίζουμε να παράσχουμε τρόφιμα, στέγη, υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας σε εκατομμύρια πληγέντες. Μάλιστα ξέχασα να αναφέρω κάτι. Δεν ξέρω ε, ποιος είναι. Έχουμε Βέλγους εδώ στην αίθουσα. Ρωτώ διότι μια ιατρική ομάδα βελγική ήταν η πρώτη που έφτασε στο Τακλομπάν για να παράσχει βοήθειας. Ε, η fast έτσι λέγεται και πράγματι ανταποκρίθηκε στο όνομα, ήταν η πρώτη. Και μια γερμανική ομάδα, η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, συλλογική δράση, ε, κατεδείχθη εκεί και πραγματικά αυτό ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για μια Ευρωπαία σαν εμένα. Συνεχίζουμε με τις ανακουφιστικές αυτές ενέργειες, δράσεις, αλλά αρχίσαμε να σχεδιάζουμε ε, πώς θα συμβάλλουμε στην ε, αποκατάσταση, ανοικοδόμηση αποκατάσταση. Θέλουμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν χρήματα και τρόφιμα για να παράσχουμε βοήθεια και να βοηθήσουμε και την τοπική οικονομία να ανακάμψει. Θέλω να εκφράσω την, την, ε, ένα θερμό ευχαριστώ στην ΔΕΦΚΟ, τη Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, προσπάθειες που έγιναν για τη σύνδεση της ε, βοήθειας για την ανακούφιση στη βοήθεια για την ανοικοδόμηση και αποκατάσταση. Και με αυτά σταματώ και για να δώσω το λόγο στον κύριο Ντεμέλο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ε, μεγάλη χαρά και τιμή που νιώθω να είμαι ενώπιόν σας για πρώτη φορά στα νέα μου καθήκοντα και επίσης να τονίσω την απόλυτη προσήλωσή μου στη συνεργασία με την Επιτροπή σας. Όπως είπε η κυρία Επίτροπος, όλα αυτά δείχνουν ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών, αλλά και μέσα στις υπηρεσίες της Κομισιόν, η ΕΦΚΟ, η ΠΕΦΚΟ, έχουν συνεργαστεί από την αρχή για να εξασφαλίσουν ότι κάθε γενική διεύθυνση με τις γνώσεις της και τις ικανότητές της θα μπορέσει να συμβάλλει στη συνολική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΦΚΟ λοιπόν και η ΠΕΦΚΟ δώσανε 10 εκατομμύρια ευρώ τα οποία μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε ο Επίτροπος Πίμπαλξ ο οποίος πήγε σε μια αποστολή προγραμματισμού στην περιοχή αυτή πήγε αμέσως στις Φιλιππίνες για να εξασφαλίσει ότι θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν η εκταμείευση των ποσών αυτών μετά την ανακοίνωση από την Επίτροπο Τζοζέβα. Έχουμε βρεθεί λοιπόν σε πολύ καλή συνεργασία και στην ε, Μανίλα και σε άλλα τμήματα του Φιλιππινέζικου Αρχιπελάγους. Το αναπτυξιακό ταμείο το οποίο διαχείριζεται η ΔΕΦΚΟ έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει την αποκατάσταση των ζημιών και την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν η ταχύτερη δυνατή και χωρίς ε, ε, ε, ασυνέχειες μεταξύ της ανακουφιστικής ανθρωπιστικής βοήθειας και της βοήθειας για ανάπτυξη και αποκατάσταση. Έχουμε ήδη ένα σχέδιο προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης από την κυβέρνηση των Φιλιππινών επί τη βάση των δικών του εκτιμήσεων των αναγκών. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν θα ακολουθήσει αυτό το πλαίσιο για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει και συμπληρωματικότητα και τήρηση των προτεραιοτήτων οι οποίες έχουν τεθεί σε εθνικό και <clears throat> διεθνές επίπεδο σε σχέση με τη χρήση των πόρων. Η ανικοδόμηση και η αποκατάσταση, οι ανάγκες για την αποκατάσταση και την ανικοδόμηση ανέρχονται κατ' εκτίμηση σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστιες αυτές οι ανάγκες. Το να γίνουν καλύτερες οι νέες κατασκευές και να αντέχουν οι νέες δομές σε φυσικές καταστροφές, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα ακόμα ποσά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως ότι η κυβέρνηση των Φιλιππινών έχει σημαντικό περιθώριο προϋπολογισμού και επομένως <clears throat> είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια ανοικοδόμησης και αποκατάσταση τα επόμενα χρόνια. Με την αντιπροσωπεία μας στη Μανίλα, εμείς είμαστε σε στενή επαφή με την κυβέρνηση των Φιλιππινών με τους εταίρους μας σε αναπτυξιακό επίπεδο και τα κρατη για να μπορέσουμε να δώσουμε την απαραίτητη βοήθεια για την ανοικοδόμηση. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό αξιολογούμε τις δυνατότητες χρησιμοποίηση των 10 εκατομμυρίων ευρώ που θα υποστηρίξουν αυτή την πρώτη φάση. Και επίσης μετά από την έλυση της τοπικής κυβέρνησης εξετάζουμε πώς μπορούν ποσά από ήδη λειτουργούν τα προγράμματα να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν την ανοικοδόμηση. Θα προσπαθήσουμε παραδείγματος χάρη να ε, επιταχύνουμε την ε, εκταμείευση ενός ποσού 10 εκατομμυρίων που προορίζεται για τον υγειονομικό τομέα και αυτό θα βοηθήσει την κυβέρνηση να ενισχύσει τις δομές υγειονομικής περίθαλψης στις περιοχές που έχουν πληγεί από τον τυφώνα. Τέλος, μέσα στα πλαίσια του προγραμματισμού για το 2014-2020 και από τη στιγμή που θα έχουμε τη νομική βάση για το DCI από τις αρχέ του προπολογισμού. Θα εξετάσουμε με την κυβέρνηση των Φιλιππινών πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα την, τις δράσεις αποκατάστασης και να βοηθήσουμε στο μέλλον τον πληθυσμό για να υπάρξει μια σωστή ανάπτυξη στους κέριους τομείς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Οι βουλευτές τώρα οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Κόρτες Λάστρα πρώτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλώς ήλθατε κυρία Επίτροπε. Εγώ σας είχα συναντήσει την προηγούμενη εβδομάδα, μιλούσαμε για τη Συρία, για την Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία και τώρα δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε την καταστροφή στις Φιλιππίνες. Είναι πολλά τα στοιχεία που μας δίνεται, αλλά βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος της βοήθειας έρχεται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές χώρες όμως δεν συμμετέχουν. Συμμετέχει σημαντικά παραγωγικά το Ρωμένο Βασίλειο, άλλες χώρες όπως και η δική μου δεν έχουν συμβάλει όσο θα έπρεπε. Έχουμε δρόμο να διατρέξουμε λοιπόν. Μίλησατε προηγουμένως για, την, ε, για το συντονισμό με τους άλλους δωρητές στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε καλύτερα πώς γίνεται αυτή η δράση συντονισμού και πώς λειτουργούν οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω και κάτι ακόμα για τις βασικές ανάγκες που έχει περιγράψει η κυβέρνηση των Φιλιππινών. Ποιες είναι οι προτεραιότητες για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί τους, τι ακριβώς ζητούν από εμά πιο κατεπηγόντως. Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα όταν μας μιλούσατε για τους πρόσφυγες στη Συρία θα ήθελα να ξέρω αν και στις Φιλιππίνες υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο και σχέδιο δράσης για τα παιδιά και τους ε, ανήλικους για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Ο κύριος ε, Μπέρμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Στρίφλα. Κυρία Επίτροπε, Είπε ακριβώ το θέλω να πω ο κύριο Λάστρα, γι' αυτό και τώρα θα πρέπει τώρα να αυτοσχεδιάσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα και για μένα. Ξέρετε, είχαμε έναν εντυπωσιακό αριθμό από εκστρατείε ε, δωρεών και οι Ευρωπαίοι παντού, παντού έχουν ε, συμβάλει γενναιόδωρα. Τι γίνεται με τον ε, συντονισμό που αφορά τη συγκεκριμένη αυτή χρηματοδότηση Πεςτε μας δύο λόγια σε αυτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, σας ξαναδίνουμε το λόγο. Επίτροπος. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Πρώτα πρώτα, για να ξεκαθαρίσουμε το ρόλο της ε, Νορβηγίας, δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής αλλά ανήκει στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Οπότε και αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα συντονισμού πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα κρατημέλη. Ας φορά τώρα τον συντονισμό με τα ε, Ηνωμένα Έθνη, πρώτα πρώτα. Θέλω να δούμε ακριβώ τι δυνατότητε έχουμε, τόσο ώστε να συντονιστούμε με τον ΟΗΕ και συνδέσαμε την ε, σε κάποια πάρα πολύ απομακρυσμένα μέρη, κάπου στο, στον ΟΗΕ και αυτό το λόγο και η κυβέρνηση των Φιλιππίνων προς τα εκεί κατευθύνει τις της και όταν πήγα εκεί εντυπωσιάστηκα που είδα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ήταν μια γροθιά. Όλοι συνεργάζονται ε, πραγματικά ενωμένα. Και αυτό γιατί πολλές φορές έχουμε κάποιες παράλληλες δομές Οπότε και χάνεται χρόνος. Στην προηγούμενη περίπτωση αυτό το οποίο έχουμε να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε με το να γίνει κάποια αξιολόγηση εκεί ε, που, χρειάζεται. Να, κοιτάξτε αυτούς τους χάρτες. Μπορείτε να ξαναβάλει το χάρτη. Για πάμε σε αυτό το χάρτη. Πρώτα πρώτα η επικέντρωση των προσπαθειών ε, στο μέρος αυτό και μετά στις γύρω περιοχέ, λόγω της μασικής χαστοδής που εκεί συνέβη είχαμε πάρα πολύ σημαντική ε, απόλυση ε, ανθρωπίνων ζωών αλλά εκεί λίγο πάνω από το Λάιτε αυτό τη, τη, πτώση όπως και το λέτε Οπότε και έχουμε και διάφορα άλλη ε, μέρη τα οποία ε, είναι πέραν πάση επικοινωνία οπότε θα πρέπει να αποκατασταθεί η κατάσταση ακριβώ όπω βοήθησε ε, επίσης στείλαμε και μια ομάδα να αξιολογήσει την κατάσταση οπότε να δούμε πόσοι χρειάζονται τρόφιμα, ε, ιατρική κάλυψη, στέγαση, στέγη κλπ. να δούμε τελικά πώς θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει. Φαίνονταν εύκολη η διαδικασία. Πάντως, από πλευράς συντονισμού των ιδιωτικών δωρεών, ε, συνήθως αυτό γίνεται ε, μέσω ε, κάποιων ε, πάρα πολύ αξιοσέβαστων ανθρωπιστικών οργανώσεων όπως η Oxfam, όπως το Save the Children, όπως το UNICEF και επίσης κατά αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε τόσο α, του ιδιωτικού τομέα. Και αυτό και πολλές φορές και εγώ σκέφτομαι πώς θα μπορέσω να καλύψω το σύνολο και να αξιοποιήσουμε αυτήν την γενοδορία. Δηλαδή να αξιοποιήσουμε για μια φορά το χρήμα των Ευρωπαίων διότι αυτές οι οργανώσεις είναι εταίροι μας, εταίροι μας στα πλαίσια του ΟΗΕ και αυτό το οποίο κάνουν ε, από τους ε, ηθιώτες τελικά είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις συλλογικές προσπάθειες. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να, ε, μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο γρηγορότερα σε κάποια μέρη. Και αυτό διότι πρόκειται για, για κάποιες επιπτώσεις που είχαν ευρεία ε, ανταπόκριση εκεί που δεν υπήρχαν επικοινωνίες. Και αυτό το οποίο έκαναν ήταν να βάλουν στις στέγες τους κάποια μηνύματα, κάποια ε, πλακάτ ζητώντας βοήθεια και περίμεναν να έρθει ε, κάποια βοήθεια δεν έχει σημασία πότε και ήρθε αλλά οι αρχές της Φιλιππίνες αλλά και εμείς ε, πήραμε το μαθημά μας ότι δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Ας πούμε είχαμε αυτές τις ε, πλημμύρες τόσο μεγάλες, αυτές που γίνανε το 2002 στην ε, το 2013 στην Κεντρική Ευρώπη αλλά θα έπρεπε να ανέβει το κατόφλι του για την ετοιμότητα. Όσον αφορά τώρα τον ορισμό των βασικών αναγκών αυτό, να δούμε τι είναι αυτό που ζητούν οι αρχές. Μιλήσαμε ε, στον ε, Υπουργό Εσωτερικών για μας ότι υπάρχει εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό πρέπει να γίνει, δηλαδή ε, πώς θα καθαρίσουμε από τα ερήπια, τα, τις αυλές των σχολείων και να γίνουν επομένω ξανά ασφαλή τα σχολεία. Για μένα αυτό απετέλεσε μια προτεραιότητα και αυτό γιατί όχι μόνο ε, κάποιες οικογένειες χάσανε τα σπίτια τους αλλά και τα παιδιά χώσαν, χάσανε το σχολείο τους, δηλαδή δεν μπορούν πια να πάνε στο σχολείο τους πέραν αυτής της ε, τρομερής τραγωδίας. Επομένως όλα αυτά τα ερήπια είναι μια προτεραιότητα. Θα είναι όλα αυτά προτεραιότητα στην ΤΕΦΚΟ. Προσπαθούμε να δούμε δύο ομάδες του είπαν προτεραιοτήτων. Απλώ ανθρωπιστική βοήθεια, πρώτα πρώτα τις άμεσες βοήθειες για την ανακούφιση αυτών των ανθρώπων, όπως αναφέρατε τα συνεργατά παιδιά, τους ανηλίκους που έχουν χάσει τους γονεί του. Ευτυχώ οι Φιλιππίνες είναι μια χώρα στην οποία έχουμε τις διευρυμένε οικογένειε και ισχύει μια τέτοια παράδοση. Οπότε η οικογένεια φροντίζει τους ηλικιωμένους, τα παιδιά κλπ. Όμως αυτό είναι και προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Το πώς οι δάσκαλοι θα ξαναγυρίσουν στα σχολεία. Επίσης, να πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους, πώς αυτοί όλοι θα είναι κορυφαία προτεραιότητα που θα την καλύψουμε. Δεν έχουμε πλέον ε, νοσοκομεία. Στο Τακλομπάν το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο ήταν ε, το, το μόνο κέντρο παροχής ιατρικής βοήθειας σε όλη αυτή την πληγήσα ε, περιοχή. Είχαμε 1.800 περίπου που κάνανε ουρά και άλλοι τόσοι ήταν μέσα στο νοσοκομείο και τους περίθαλπους η ΔΕΦΚΟ επομένω θεωρήσε ότι αυτά είναι προτεραιότητα και εμεί το θεωρήσαμε ότι έτσι έχουν τα πράγματα για να δούμε πώ θα υπάρχει άμεση ενίσχυση και πώ θα έχουμε το δεύτερο πακέτο, δηλαδή το πώ θα βοηθήσουμε την συγκρότηση, πώ η ανθρωπιστική βοήθεια θα χρησιμοποιηθεί για να ξαναδημιουργήσει θέσει από για τον κόσμο, να καθαρίσουμε τα σχολεία από τα ερήπια. Αυτό είναι μια κλασική κίνηση από όλοι βγαίνουν κερδισμένοι, να δούμε τι γίνεται με αυτούς που χάσαν τις δουλειές τους, γιατί βρήκαμε ε, κάποιους χώρους ασφαλείς για τα παιδιά, εκεί που ε, είχαμε ε, πάρα πολλές φορές συνέπειες καταστροφής και να, θέλουμε να δούμε πώς θα γίνει η επιστροφή, γιατί εκτός από του τους ανηλίκους Οφείλθηκαν και οι ενήλικες και οι γονείς, γιατί κάπου συνειδητοποίησαν ότι η ζωή ξαναπεί τους φυσιολογικούς ρυθμούς. Α, κάτι άλλο, εάν μου επιτρέπετε, σε σχέση με τις ανακοινώσεις της ε, κυβέρνησης, ε, ήρθε σε επαφή μαζί μου ο ή υπουργός εξωτεριών. Ε, πρόκειτο περί εκφράσης γνωμοσύνης για όσα έκανε η Ευρώπη. Επίσης ε, το, ίδιο ένα πολύ πολύ θερμό ευχαριστώ από την Βουλή της χώρας. Αλλά πιο πολύ θερμά ευχαρίστησαν οι άντρε και οι γυναίκε που στα νοσοκομεία και που όλοι αυτοί είπαν μια φωνή. Ευχαριστούμε πρώτα για όσα έκανε για μα. Η πρόεδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σβέντσον, θέλετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για την αφοσίωσή σας και για την ε, παρουσίαση την ενθαρρυντική για το τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που μπόρεσε τόσο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσει στις Φιλιππίνες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλό είναι να ακούσαμε και για τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένες Πολιτείες, ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς στείλαμε μεγάλα ε, κοντέινερ και με τα πλοία έφτασαν γρήγορα. Η Ιαπωνία και η Κίνα, ξέρετε να μας πείτε τι έκαναν και εκείνες για να βοηθήσουν τις Φιλιππίνες. Εμείς ε, είχαμε επαφή με τους εταίρους μας στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Εκείνοι έδωσαν και στρατιωτικές ε, δυνατότητες πολύ χρήσιμες. Επίσης η Ιταλία τώρα συμμετέχει με το στρατιωτικό νοσοκομείο στην περιοχή. Επίσης ε, παράσχαμε ε, στρατιωτικές δυνατότητες πολύ σημαντικές και ενώ βελτιώνουμε την ορατότητα της δράσης μας ως Ευρώπη, οι Αμερικανοί φίλοι είναι πιο αποτελεσματική στην περιοχή. Δηλαδή ακόμα εμείς έχουμε πολλά να μάθουμε. Ο κύριος Κόρτες στο τέλος είπε πολύ σωστά ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία είναι οι πιο γενναιόδορες ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά εκεί. Επίσης, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ε, κάποια μικρή βοήθεια σε είδος από την Ευρώπη ήταν το ίδιο πολύτιμη, αν όχι και πολύτιμότερη, λόγω της έγκαιρης άφηξής της σε απομακρυσμένες περιοχές. Δεν πρέπει να υποτιμάμε αυτό που κάναμε. Καμιά φορά μπορεί να είναι μικρή βοήθεια, αλλά αν είναι στοχευμένη και έγκαιρη, είναι πολύ πιο σημαντική για τους πληγέντες από ότι η μεγάλης κλίμακας βοήθεια στις ε, πλέον πληγήσεις περιοχές. Τώρα για την Ιαπωνία και την Κίνα. Εγώ έτυχε να είμαι στην ε, Ιαπωνία όταν χτύπησε ο τυφώνας. Είχαμε με Ιάπωνες ε, συναντήσεις συντονιστικές. Μετά πήγα στην Κίνα γιατί ήταν ο επόμενος προορισμός μου. Στην αρχή υπήρχε στην Κίνα κάποια απροθυμία για ανάληψη δράσης, κυρίως επειδή και εκείνοι επλήγησαν από τον τυφώνα Χαγιάν. Ε, Κατομμύρια άνθρωποι ε, Κινέζοι επλήγησαν από τον τυφώνα Χαγιάν. Όμως ε, μετά από κριτική που τους έγινε αύξησαν την συνεισφορά τους. Αυτό που ήταν κέρια σημασία είναι ότι στις Φιλιππίνες ο συντονισμός των δραστηριοτήτων από, από τον ΟΗΕ και τις Φιλιππινέζικες αρχές και βεβαίως με τη δική μας συμβολή του, του δικού μας προσωπικού βοήθησε στην ε, πιο ισομερή κατανομή της βοήθειας. Αυτό έγινε με καλύτερο τρόπο από ό,τι άλλες φορές. Και ε, ανέφερα και το ε, μηχανισμό πολιτικής ε, προστασίας και πώς δημιουργήθηκε μετά το σεισμό στην Τουρκία ε, δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός όπου στείλαμε πολλή βοήθεια, πολλές ομάδες και μετά διαπιστώσαμε επικαλύψεις δεν υπήρχε συντονισμός και πήγαιναν στα ίδια σπίτια δύο και τρεις φορές. Τώρα αρχίζουμε να συντονιζόμαστε και περηφανεύομαι που μπορώ να πω ότι σε αυτή την περίπτωση καταδείξαμε την αξία του συντονισμού, γιατί σώθηκαν περισσότερες ζωές σε τελευταία ανάλυση και βοηθήθηκαν περισσότεροι άνθρωποι ε, την τραγική εκείνη στιγμή. Θέλετε να λάβετε και εσείς το λόγο κυρία Γενική Διευθυντά. Δεν είναι πολύ. Ναι, ναι, πρέπει να σας πω ότι βεβαίω και με άλλους νόμους συνεργαζόμεθα και με την Παγκοσμία Τράπεζα και με την Ασιατική Τράπεζα. Οπότε και γι' αυτό και θέλουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φασίσουμε για ε, το δάνειο. Ε, χρειάζεται αυτό να γίνει και σε αυτό το επίπεδο. Κύριε Νάιζερ, θέλετε το λόγο. Να ευχαριστήσω και εγώ πολύ την Επίτροπο Αναφερθήκατε στο μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Βλέποντας τον κατάλογο και την οικονομική συνεισφορά των επιμέρους κρατών μελών, βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Οι οικονομικά ισχυρές χώρες είναι μια κατηγορία, οι λιγότερο ε, ισχυρές οικονομικά χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε έναν μηχανισμό που θα ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες των χωρών. Δύο παραδείγματα. Η Μεγάλη Βρετανία έχει 66 εκατομμύρια ε, ευρώ βοήθεια. Η Γερμανία δίνει το 1 δέκατο. Αυτά τα 6 εκατομμύρια της Γερμανίας καλά είναι και αυτά. Αλλά σε σύγκριση με το, ότι το Ηνωμένο Βασιλείο είναι μια πενιχρή συνεισφορά από μια χώρα που είναι οικονομικά ισχυρότερη. Και υπάρχουν και άλλες ανισότητες. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό αν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα ε, γινόταν μια προσπάθεια για καλύτερη ισορροπία σε σχέση με την οικονομική ευρωστία κάθε χώρας. Βεβαίως ε, κάθε χώρα μπορεί να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με μια χώρα που πλήττεται από καταστροφή. Αλλά όταν συντονίζεται η βοήθεια μεταξύ των κρατών μελών, η ευρωπαϊκή βοήθεια, η ενωσιακή βοήθεια, ε, νομίζω ότι δεν πρέπει, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν τέτοιες διαφορές μεταξύ οικονομικά ισχυρών και λιγότερο ισχυρών. Δεν επιτρέπονται τέτοιες ανισότητες όπως αυτές που βλέπουμε σε αυτό τον κατάλογο πάρα πολύ μεστές αυτές οι σκέψεις. Θα θέλατε να απαντήσετε, κύριε Επίτροπος. Πρόκειται για ιστορία που έχει ακόμα μέλλον όσον αφορά τις δυνατότητες να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προσοχή κύριε μέλλον; Μιλάμε για 1,7 δις ευρώ ζημίες. Άρα, εδώ έχουμε πολύ περιθώριο συμβολής και βοήθειας προς τον πρώτο μελών. Τέτοιο είδους δεν μπορεί να γίνει. Πάντως δεν θα είναι αυτό το τέλος των προηγούμενων προσπαθειών. Είπαμε να γίνει μια διάσκεψη, ούτω ώστε να υπάρξει βοήθεια προς τη χώρα κάποια στιγμή αργά τέλη Δεκεμβρίου. Οπότε και έτσι να βρεθούν κάποια ευκαιρία για ποιε χώρε οι οποίε έχουν περισσότερε δυνατότητε, ούτω ώστε να αναλάβουν δράση επ' αυτού. Έχετε δίκιο, έχουμε και άλλα θέματα εδώ και η Γερμανία είναι αλήθεια ότι ε, βέβαια τα 6,6 εκατομμύρια αποτελεί έκφραση γενετορία σε σχέση με το ότι το Ηνωμένο λιγότερο. Πάντω έλεγα ότι όσον αφορά τη Συρία, η Γερμανία ε, ε, κάνει πολλά, κάνει, επιτελεί πάρα πολύ σημαντικό έργο και οικονομικά η συμφωνία της Γερμανίας είναι πάρα πολύ βαρύνουσα. Τώρα υπάρχει κάτι το οποίο ω αρμόδιο επίτροπος με ενοχλεί, με απασχολεί το να δούμε το κατά δεν θα ξεχαστεί καμία κρίση. Είπαμε και την κεντροφυγική δημοκρατία εδώ τις προάλλες. Ε, θεωρούν αυτούς χώρα ξεχασμένη άρα. Αυτό θα πράγμα. Άρα έχετε δίκιο. Θα υπάρχει περιθώριο να μπορέσουν να ζοριστούν κάποιοι κρατημένοι και να κάνουν λίγο παραπάνω. Κορτές Λάστρα. Μια άλλη ερώτηση κυρία Επιτροπέ. Ναι, είπατε ότι προσωστερικών κλπ. Και είδαμε σε μια σειρά αποστολών ε, που ανέλαβε η Επιτροπή Ανάπτυξης, είδαμε τι γίνεται όσον αφορά το πόσο μπορούμε να συντονιστούμε σαν αντιπροσωπείε, σαν πρεσβείες. Βέβαια εδώ πέρα ήταν τι εξελίξεις, με ξεπέρασαν με ένα σημείο, εσείς βέβαια ξέρετε. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αυτή η υπόθεση. Υπάρχουν κάποιε χώρε οι οποίε δεν είναι πολλά και κατά κάποιο τρόπο είναι διαθέσιμε. Όμω θα πρέπει όλη αυτή η βοήθεια να συντονίζεται και δεν είναι δυνατόν ο καθένα να κάνει ό,τι του έρχεται. Σύμφωνοι, κάθε βοήθεια τώρα είναι απαραίτητη. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Τι είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο του Φιλιππινέζου. Και έτσι και εμεί να κάνουμε τα αντίστοιχα, τα ανάλογα. Άρα να δούμε πώς λειτουργήσε αυτή, αυτός ο συντονισμός. Μπορέσουμε να συντονιστούμε. Δουλέψαμε με τον πιο δόκιμο τρόπο. Αυτό αν κάνουμε τότε θα είμαστε όσο είναι πιο αποτελεσματικοί και πιο χρήσιμοι για τις Φιλιππίνες. Τελευταία ερώτηση. Απαντήστε. Ε, είμαστε πολύ υποχρεωμένοι και ευγνώμονες προς τον πρέσβη μας και την αντιπροσωπεία μας στη Μανίλα που δούλεψαν 24 ώρες επί 7 μέρες τη βδομάδα για να δοθεί σωστά η βοήθεια. Εμείς έχουμε περιφερειακά γραφεία κοντά σε περιοχές που είναι πιθανόν να υπάρχει, ε, να υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή των ομάδων στη Μπαγκόγκ και βεβαίως ε, αντέδρασαν ανάμεσα. Έχουμε ένα μικρό γραφείο στις Φιλιππίνες. Τώρα υπάρχει μόνιμη αντιπροσωπεία για τους επόμενους 6 ε, με 12 μήνες, ανάλογα με το πόσο θα διαρκέσει η δράση μας εκεί. Και είχαμε τις δύο ομάδες, ανθρωπιστική ομάδα και την ομάδα πολιτικής προστασίας που δούλεψαν ως μία. Η απόφαση συγκερασμού των δύο ομάδων σε μια υπηρεσία, ανθρωπιστική και πολιτική προστασία, απεδείχθη σωστή απόφαση γιατί μπορέσαμε έτσι να αναβαθμίσουμε τις ε, ικανότητές μας ε, εκτίμησης της κατάστασης και για να δούμε πάλι στη διαφάνεια, πίσω πηγαίνετε για να δούμε τις ομάδες αξιολόγησης και εκτίμησης της κατάστασης. Βλέπετε εδώ τα μέλη της ομάδας εκτίμησης, είτε είναι ειδικοί για την ε, ε, ανθρωπιστική βοήθεια ή για την πολιτική προστασία, είτε από τα κράτη-μέλη ειδικοί, είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έδρασαν όλοι μαζί. Και έτσι μπορέσαμε, τολμώ να πω, στην καλύτερη δυνατότητα εκτίμησης της κατάστασης και συμβάλαμε και στην εκτίμηση που έγινε από τα Ηνωμένα Έθνη. Ακριβώς επειδή είμαστε τώρα οργανωμένοι έτσι, έχουμε μεγάλη ευελιξία ανάπτυξης ε, ικανοτήτων. Έχουμε τρεις πυλώνες. Τη ε, περιφερειακή δράση του ΕΚΟ, την ομάδα πολιτικής προστασίας συνδεδεμένη με την ομάδα ε, την ανθρωπιστική για φυσικές καταστροφές και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και τις ικανότητες των κρατών μελών. Δηλαδή, κάποια κράτη-μέλη είχαν τις δικές τους ομάδες εκτίμησης της κατάστασης. Τώρα λειτουργούν σε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο. Έτσι έχουμε πολύ καλύτερη στόχευση και πιάνει τόπο το κάθε ευρώ σε ό,τι αφορά δηλαδή τα ωφέλη που θα δώσουμε στους πληγέντες. Δεν θέλετε. Ο Γενικός Διευθυντής δεν θα ζήτη το λόγο. Κυρία Γεώργιεβα, σας ευχαριστώ. Κύριε Φουτού, όσο δεν μέλλον επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και μας δώσατε μια εκτίμηση της κατάστασης στις Φιλιππίνες χαίρομαι πάρα πολύ που μπορείτε να κάνετε όλα αυτά τα οποία είναι ανθρωπίνως εφικτά για να μπορέσει να αναπτυχθεί η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και να γίνει αποκατάσταση στα πρώτα στάδια τουλάχιστον στις Φιλιππίνες. Σας ευχαριστώ πολύ, έρχεστε πολύ συχνά εδώ και είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.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 Λοιπόν, όπως θέλετε ακριβώς. Για το επόμενο μας σημείο της ημερησίας διάταξης έχουμε τη μεγάλη τιμή να υποδεχθούμε τον κύριο Ζερεμι Λεφρούα από το, τη Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ελλονοσία και τις παραμελημένες τροπικές ασθένειες και τον κύριο Σεμπερκλέ, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής της Gavi Alliance. Με την παρουσία τους θα μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερο για την πρωτοβουλία κατά των ασθενειών που αφορούν ιδιαίτερα και δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο κύριος Ζεφρόα ήταν επικεφαλής μια ομάδα που έχει εκπονήσει μια έκθεση για την Ελλονοσία και ο κύριος Μπερκλέη θα μας παρουσιάσει <clears throat> τις δράσεις της ε, οργάνωσής του για τον εμβολιασμό των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της κατάστασης για τις ασθένειες που συνδέονται με την ένδια. Παραμένει όμως πολλής δρόμος να διατρέξουμε και πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ξέρουμε ότι 600.000 άτομα, κυρίω παιδιά, πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω ελανοησίας και 1,7 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειε, οι οποίε θα μπορούσαν να, να, προληφθούν συγγνώμη, με την εμβολιασμό. Δίνω το λόγο στου ε, καλεσμένου μα για 10 λεπτά τον καθένα και μετά ζητώ από του συναδέλφου να λάβουν το λόγο και να θέσουν κ. Λεφρουά για 10 λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Η Επιτροπή μας στο Κοινοβούλιο ε, του Ηνωμένου Βασιλείου σας έχει στείλει την έκθεσή μας για την Ελλονοσία του 2013 και επίσης δημοσίευσαν την προηγούμενη εβδομάδα την έκθεσή μας για τις ε, παραμελημένες ασθένειες και θα σας αφήσω και περαιτέρω αντίγραφα. Η έκθεσή μας για την Ελλονοσία με τίτλο «Η Ελλονοσία στο Σταυροδρόμι» έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας. Πολλά έχουν γίνει εναντίον της Ελλονοσίας από τότε που άρχισε μια σοβαρή αντιμετώπιση της πριν από 10 χρόνια περίπου. Αλλά εάν συνέχιζε η θνησιμότητα που ίσχυε το 2000 θα είχαμε 274 θανάτους θα είχαμε 274.000 παραπερισσότερους θανάτους. Έχει μειωθεί λοιπόν ε, σημαντικά η ελονοσία και θέλουμε μέχρι το 2015 να μειώσουμε τα κρούσματα ελονοσίας κατά 75% έναντι του 2000. Υπήρξε μεγάλη πρόοδος για την διανομή και τη χρήση εντομοκτώνων κατά του ανοφελούς κόνοπο, κόνοπος σε περισσότερα ε, τεστ και δοκιμασίες και στη χρήση περισσότερων φαρμάκων σε συνδυασμένες θεραπείες. Βλέπουμε μεγάλη ε, πρόοδο με την χρήση νέων εμβολίων και έχουμε λοιπόν μια καλύτερη εργαλειοθήκη από ό,τι είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη, είτε πολυμερό είτε διμερό, μέσω του συνολικού ταμείου, οργανώσεων όπω η Γάβη κτλ., ήταν κεφαλαιώδη για την επίτευξη των στόχων μα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη έχει παίξει σημαντικό ρόλο και χαιρετίζω τι προτάσει για ένα νέο τέτοιο αναπτυξιακό ταμείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε όμω τι προσπαθίε μα. Έχω ζήσει 11 χρόνια στην Τανζανία και στη δεκαετία του 50 και του 60 λεγόταν ότι είχε εξαλειφθεί η ελονοσία από τη Ταρσία τη Ανζιβάρης αλλά επανερχόταν κάθε φορά που σταματούσαν οι προσπαθίες μα. Έχω δει πολλού φίλου μου να πλήττονται από αυτήν την ασθένεια και εγώ ίδιο έχω περάσει ελονοσία. Στην αρχή είχα ένα, πήρα ένα φάρμακο που λεγόταν Λάριουμ και είχε πολλές παρενέργειες. Μετά πήρα νέα φάρμακα και είδα πόσο βελτιώνεται η κατάσταση με τα νέα φάρμακα τα οποία δεν έχουν παρενέργειες. Γι' αυτό έχω επενδύσει μαζί με πολλούς φίλους τις προσπάθειες για να αναπτυχθεί η χρήση των νέων φαρμάκων. Δεν είχαμε όμως αρκετά χρήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη και πεθαίνανε χωρίς λόγο άτομα παρά το γεγονός ότι υπήρχαν τα απαραίτητα φάρμακα. Θέλω να τονίσω ότι χάσαμε πάρα πολύ χρόνο από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι το 2000. Αν ήταν ασθένειες στις δυτικές χώρες δεν θα είχε γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια σφάλματα. Πρέπει να αναπτύξουμε διαγνωστικές μεθόδους, προληπτικές μεθόδους και εμβόλια για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και τώρα έχουμε δύο ε, μορφές ε, ελονοσίας στην Νοτιοανατολική Ασία που αντέχουν στην Αρτεμισία και όπως ξέρετε υπάρχουν και μορφές που, που δεν αντιμετωπίζονται με το Chloroquine που ήταν το πρώτο φάρμακο που ήταν πραγματικά αποτελεσματικό και τώρα βρίσκονται αυτές οι μορφές στην Αφρική και στην Ινδία. Μια ε, ομάδα πήγε στη Μιανμάρ εκεί πρόσφατα και είπε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Χρειάζεται τώρα να αναχαιριστεί η εξάπλωση της ελονοσίας. 100 εκατομμύρια δολάρια είναι τα συνολικά ποσά που έχουμε στη διάθεσή μας, χρειάζονται όμως περισσότερες προσπάθειες για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες. Ναι, η πρόεδρο ζητάει να μειώσει την ταχύτητα του ομιλητή για του διερμηνείς. Έχουμε λοιπόν σημαντικές ε, προσπάθειες, αλλά υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι αν δεν μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα φάρμακα. Επίσης η δεύτερη αντιμετώπιση είναι τα εντομοκτώνα σε κουνουπιέρες για να σκοτώνουν τα έντομα. Αυτά, αυτές οι κρουπιέρες οι οποίες έχουν εμποτιστεί με φάρμακα κατά των κονόπων είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο κατά της ελονοσίας. Αν όμως σταματήσει να είναι αποτελεσματικό αυτό το δίκτυ, τότε η κουνουπιέρα τότε δεν μπορεί να προστατεύσει. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, διότι στις χώρες που έχουν το μεγαλύτερο βάρος λόγω αυτής της ασθένειας. Οι 14 χώρες αυτές καλύπτουν τα 80% όλων των θανάτων μετά από τις μεγάλες προόδους της τελευταίας δεκαετίας βλέπουμε να μειώνεται ο ρυθμός της προόδου. Η χρήση των κουνουπιερών ήταν 3% το 2000 και είναι 53% το 2011 αλλά δεν έχει αυξηθεί το 2012. Η ετήσια έκθεση για την Ελλονσία του 2012 εκφράζει ανησυχίες ότι μπορεί να έχει φτάσει σε ένα σημείο τελμάτωσης η χρήση αυτής της, ε, των κουρουπιερών τη στιγμή που δεν υπάρχει περαιτέρω χρηματοδότηση. Έχουμε την ανάγκη να φτάσουμε στο 1,5 δισεκατομμύρια το χρόνο μέχρι το 2020 για να μπορέσουμε να έχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2,5 ε, εκατομμύρια, 1,8 από διεθνούς οργανισμούς και 600 περίπου χιλιάδες από, εθνικές, από εθνικούς πόρους. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αυξηθούν οι πόροι αυτοί και να υπάρχουν και περαιτέρω δωρητές. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξήσει σε ένα δισεκατομμύριο λίρες μέσα σε τρία χρόνια τη χρηματοδότησή του και αυτό είναι τμήμα της δέσμευσης του Ηνωμένου Βασιλείου για να αυξηθεί σε 500 εκατομμύρια λίρες η χρηματοδότηση μέχρι το 2015 μόνο για την Ελλονοσία. Τονίζουμε όμως ότι οι κυβερνήσεις των χωρών όπου είναι ενδημικές αυτές οι αρρώστιες πρέπει να τηρήσουν την υπόσχεση που έχουν να δαπανίσουν 15% του εθνικού του προπολογισμού για την υγεία. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί καλύτερα η αλλοσία και άλλε ασθένειες. Μερικέ φορέ το πέτυχαν. 80% όμω δεν το έχουν κάνει και 40% από όλε αυτέ είναι κάτω από το 10% στον προπολογισμό του. Πιστεύουμε ότι οι ιδιωτικοί φορεί και τα ιδρύματα μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Εμεί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη του εμβολίου RTSS και το γεγονό ότι μεγάλε φαρμακευτικέ εταιρείε έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα να αναπτυχθούν φάρμακα για τροπικέ ασθένειε, όπω τονίζει και η εκθέσή μα. Αλλά αυτή τη στιγμή με το περιορισμένο τμήμα του ΑΕΠ που αποδίδεται στα θέματα αυτά πρέπει ο ιδιωτικό τομέα να κάνει παραπάνω. Επομένω, το Συμβούλιο και η Κομισιόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω προχωρούμε στο δεύτερο EDC, είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι κάτι πολύ θετικό. Μόνο με τι κλινικέ μελέτε και τι δοκιμασίε μπορούν οι χώρε μα να βοηθήσουν στα θέματα αυτά. Με το να εξασφαλίσουν ότι οι νέε αυτέ θεραπείες μπορούν να περάσουν μια ταχεία διαδικασία επαλήτευσης και έγκρισης και δεύτερο με το συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε χώρες όπου ενδημούν αυτές οι ασθένειες για να βελτιώσουμε τις ερευνητικές τους ικανότητες και τα μέσα τα οποία προτείνουμε, ιδίω η συνεργασία με άλλους μεγάλους δημόσιους και ιδιωτικούς χορηγούς μεταξύ των οποίων και οι φαρμακευτικές βιομηχανίες θα βοηθήσουν περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Στα χρόνια αυτά που ήμουν επικεφαλή αυτή τη ομάδα, αυτό που μου έδωσε τη μεγαλύτερη χαρά και ενθουσιασμό για την αντιμετώπιση τη ε, ελονοσία και άλλων ασθενειών είναι η συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, ερευνητικών φορέων, ε, ΜΚΟ και του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξαλείψουμε την ολομέλεια, την, ε, συγγνώμη, την ελονοσία και τι περισσότερε παραμελημένε ασθένειε. Δεν πρέπει λοιπόν να χαλαρώσουμε τι προσπάθειέ μα. Ευχαριστώ. Η ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπέρκλι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη συμπληρωματικότητα μεταξύ διμερού υποστήριξη και πολυμερού, όταν πρόκειται για εμβολιασμού και συστήματα υγεία και η Κομισιόν ε, τώρα ε, είναι υπεύθυνη ε, για, στο Συμβούλιο της Γκάβη και ε, θέλουμε να αναβαθμίσουμε την παρέμβασή μας όπως είπε και ο Επίτροπος. Επίσης ε, ε, χαίρομαι που το πρόγραμμα EDCTP ξαναμπήκε στην μερίσια διάταξη. Για όσους δεν γνωρίζουν την ΓΑΒΗ, υπάρχουν τέσσερις βασικές στρατηγικές. Ο στόχος του εμβολιασμού είναι ο πρώτος, δηλαδή νέα εμβόλια για αυτούς που τα χρειάζονται στις πτωχές χώρες. Ενίσχυση της υγείας είναι το δεύτερο. Το τρίτο αφορά την, ε, τα οικονομικά, ούτως ώστε να υπάρχει ε, βιώσιμη χρηματοδότηση και το άλλο είναι η διαμόρφωση της αγοράς. Θα σας ε, τα δείξω όλα αυτά σύντομα στην παρουσίασή μου. Εδώ έχουμε ένα νέο εμβόλιο. Βλέπετε εδώ την εξάπλωσή του στον κόσμο ε, παρουσιάζεται ως νέο εμβόλιο το 501 ε, υπάρχει στις, ε, σε όλες τις φτωχές χώρες με την εξαίρεση του Νότιου Σουδάν που δεν υπήρχε όταν άρχισε η δράση της Ιγκάβη αλλά στις αρχές του 2014 θα πάει το εμβόλιο και εκεί θα έχουμε ε, κάλυψη όλων των χωρών. Τώρα, για πρώτη φορά βλέπουμε μια κίνηση, βλέπετε εδώ υψηλού εισοδήματος χώρες, ε, δεξιά χαμηλού εισοδήματος και εδώ ε, μιλάμε για ισότητα, δηλαδή τα ισχυρά εμβόλια πρέπει να πάνε στις φτωχές χώρες. Και βλέπετε ότι οι περισσότεροι, ε, τα περισσότερα κρούσματα υπατήτηδας Β είναι στις χαμηλού εισοδήματος και το, επίσης το ίδιο ισχύει για τον αιμόφυλο και την γρήπη 2. Εδώ ε, από την καλύφη στην Κένια, μια διαφάνεια, ε, βλέπουμε εξαφάνιση, εξάλληψη της νόσου. Αυτό είναι το συγκλονιστικό αποτέλεσμα του εμβολίου. Τώρα ε, επιταχύνουμε πάρα πολύ. Πάμε στο NGD4 που θα, έχει, θα, επιτελέσει, θα σημάνει μεγάλη πρόοδο. Ε, εδώ η ενάρξη εμβολιασμών, ε, εξέλιξή τους διαχρονικά. Τελευταία το Συμβούλιο ε, συμπεριέλαβε το IPV ως εμβολιασμό ρουτίνας για την ε, πολιομιλίτιδα και βλέπετε ε, ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση του έργου της Gavi Alliance. Η Λαρά, σημαντική προτεραιότητα και εδώ στην Ευρώπη όπου συνεχίζουμε να βλέπουμε επιδημίες της νόσου σε διάφορες περιοχές και της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Βλέπετε εδώ τα αποτελέσματα του εμβολιασμού για η ΛΑΡΑ σε περιοχές νότιες ούτως ώστε να έχουμε όχι μόνο το εμβόλιο αλλά και μια δόση που θα διεγείρει το νοσοποιητικό. Επίσης τώρα έχουμε για την, την ερυθρά ε, εμβόλιο το οποίο επηρεάζει και τις κοίησεις πολλές φορές. Ένα άλλο σημαντικό είναι η σύγχυση μεταξύ λιμόδου, νοσού και μη μεταδοτικού. Ε, γνωρίζομαι το ε, θάνατο ε, νεαρών μητέρων ε, με πολλά νεαρά θύματα. Εδώ αντιμετωπίζει το πρόβλημα το εμβόλιο. Μειώνονται τώρα οι θάνατοι των νεαρών μητέρων αλλά αυξάνεται ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας. Περισσότεροι θάνατοι οφείλονται σε αυτό παρά στο θάνατο κατά τη γέννα. Τώρα υπάρχει εμβόλιο κατά του, τραχύλου, του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και προσπαθούμε να το διαθέσουμε τους κατοίκους των αναπτυσσομένων χωρών. Ε, η Γκάβη λοιπόν θέλει να εμβολιάσει 243 εκατομμύρια παιδιά επιπροσθέτως και είχαμε την ενδιάμεση αξιολόγησή μας και βλέπουμε ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται. Ε, τώρα, για να το δούμε προοπτικά, από το 2011 μέχρι το 2015 εμείς ε, κάναμε τους μισούς εμβολιασμού στον κόσμο, δηλαδή εμβολιάσαμε τα μισά παιδιά ε, στον κόσμο και αυτό οδηγεί σε διάσωση 4 εκατομμυρίων ζωών. Η Γκάβη τώρα λοιπόν ε, βλέπουμε ότι ε, ε, λειτουργεί σε μεγάλη κλίμακα, 250 εκατομμύρια είδαμε άλλα εκστρατείες 250 εκατομμύρια για εμβολιασμού, 400 σε εκστρατείε, ώστε να αυξήσουμε τον αριθμό των ε, ζώων που σώθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ε, δεν προλαμβάνουμε μόνο την νόσο, επηρεάζομαι και θετικά επίσης την οικονομία. Βλέπετε κάποια στατιστικά στοιχεία ει ό,τι αφορά τα περιστατικά που αποτρέψαμε και το κόστος που εξοικονομήσαμε σε σχέση με την νόσο. Πολύ μεγάλα νούμερα τα οποία δείχνουν το ενισχύ και την εξοικονομητική επίπτωση των εμβολίων. Πώς τα καταφέραμε. Έχουμε τρεις τρόπους για να συνεργαστούμε σε ένα ενάρετο τρίγωνο ε, με χρηματοδότηση από δωρητές, από χώρες και διαμόρφωση αγοράς. Η Κομισιόν βέβαια συμβάλλει, ε, συνέβαλε ε, όλο αυτό το διάστημα ε, στο 1% των κονδυλίων κάποιου προέρχονται από την Κομισιόν. Ε, και οι χώρες συμβάλλουν δεν υπάρχει πολιτική και όφελος δωρεάν, θα πρέπει να καλυφθούν από χώρες τα, το κόστος των εμβολίων ανάλογα με την οικονομική ισχύ της χώρας. Και βλέπετε εδώ αυξανόμενο ποσοστό συνεισφορών από ε, δύο ε, δεν συνέβαλαν, τώρα όμως ε, έχουν δώσει τα οφειλόμενα αν θέλετε και αυτό είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν και ευάλωτες χώρες ή χώρες που τώρα προσπαθούν να εξηγιάνουν τους προϋπολογισμούς. Διαμόρφωση αγοράς, πολύ σημαντικό στοιχείο. Ε, με μεγάλη επίπτωση γιατί εμείς ε, δίνουμε εμβόλια για στο 65% ε, της ομάδας των γεννήσεων και έτσι προσεγγίζομαι τα στοιχεία για ολόκληρο τον κόσμο και τις στατιστικές της ΠΟΗ. Εμείς σκεφτόμαστε βεβαίως όχι μόνο την συνεισφορά της ΓΚΑΒΗ αλλά τη συνεισφορά σε όλες τις χώρες. Επίσης μειώσαμε κατά 90% το κόστος για τη Δύση. Αυτό είναι σημαντικό για τη μακροπρόθεσμη ε, βιωσιμότητα των προγραμμάτων των χωρών καθώς ε, ε, έχουν, οι χώρες φεύγουν από την κάθε το, το, το κόστος ε, ήταν μεγαλύτερο στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, αλλά αφήστε με να τελειώσω. Η Γκάβη ε, αξιολογήθηκε και από τη Σουηδία το Ηνωμένο Βασίλειο βλέπετε την αξιολόγηση βαθμολογηθήκαμε καλά επίσης είμαστε στην διεθνή διαφάνεια που μας ε, έβαλε νούμερο 2 στον κόσμο για τη δουλειά που κάνουμε. Βλέπετε εδώ μεγάλο ε, βαθμό αλλά δεν είναι ολαρόδινα. Ένα κρίσιμο θέμα που μας απασχόλησε αφορά την ισοτιμία των χωρών, την ισότητα. Η Ρουάντα ε, παρουσιάζεται εδώ, βλέπετε εδώ ε, το, το ιδεώδεσε Η Νιγηρία έχει μεγάλες διαφορές, δεν υπάρχει καλή κάλυψη για όλους παρόλο που οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Τέλος, ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο εμβολιασμό έχει επιτυχία. Αν ρωτήσετε ποιο ποσοστό των παιδιών στον κόσμο ε, έχουν κάνει τα 11 εμβόλια που ε, συστήνει η ΠΟΗ, είναι 5% περίπου. Και όπως βλέπετε μέχρι το 2020 ελπίζομαι να έχουμε ε, εμβολιασμένα παιδιά στο μισό της χώρας. Όμως οι φιλοδοξίες μας είναι μεγαλύτερες. Θέλουμε αυτά τα εργαλεία να φάσουν στον καθένα που τα χρειάζεται. Τέλος να πω ότι στην προηγούμενη περίοδο εμβολιάσαμε 243 ε, εκατομμύρια και ε, προλάβαμε 400 εκατομμύρια θανάτων την επόμενη περίοδο που επεξεργαζόμαστε τώρα τη στρατηγική θα εμβολιάσουμε περισσότερα παιδιά κατά 24% και θα έχουμε ε, προλήψει θανάτων στο, σε περισσότερο από 50% των κρουσμάτων. Σταματώ και θα χαρώ να απαντήσω σε ερωτήσεις. Η πρόεδρο ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο λόγο ει του βουλευτά. Παρακαλώ. Να πείτε ποιον θέλετε να ερωτήσετε. Κύριε Γκέρτσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους δύο προσκεκλημένους μας, οι οποίοι με τις παρεμβάσεις τους μας είπαν μια πάρα πολύ επαγγελματική έποψη των πραγμάτων και Επίσης θα πρέπει να συγχαρούμε το Ηνωμένο Βασίλειο για το έργο του όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια γενικότερα. Το παραλαμβάνω συνεχώς είναι μία από τις λίγες που στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τη μία χρονιά μετά την άλλη αυξάνει την αναπτυξιακή βοήθεια. Αξίζει αυτό να το τονίζουμε και να τον αδεικνύουμε τέλος πάντων ε, εμείς έχουμε την κρίση των δύο ε, προσδεκτημένων μας, και να μας πούν την απάντηση στην πρώτη ερώτηση που αφορά το τι ισχύει όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία στα πλαίσια του ΠΟΕ. Μπορείτε να μου πείτε με κάποια ακρίβεια το τι ισχύει όσον αφορά τις επιπτώσεις των όσων κανόνων εφαρμόζει ο ΠΟΕ. έχετε προσκλούσει σε εμπόδια όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν ε, τα εμβόλια για τις αντισόμενες χώρες. Σε ποιε περιπτώσει ε, ισχύει κάτι τέτοιο, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ο ΠΟΕ πολλέ φορέ αδίκω ή δικαίω θεωρείται ένα φραγμό στην ψυχική ε, βοήθεια. Δεύτερη ερώτηση. Είχε να κάνει με τους δωρητές του ιδιωτικού τομέα, όπως το Ίδρυμα Bill Gates που έχει αναπτύξει δραστηριότητα στα πλαίσια δραστηριοτήτων που περιγράψατε. Ο ίδιος ο Bill Gates δύο φορές ήρθε εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι εντυπωσιακή η δράση που έχει αναπτύξει. Οπότε το το εξή, μια που έχουμε κάποιους θεσμικούς δωρητές. Υποστηρίζονται από τα κράτη, από τα κοινοβούλια, κοινοβούλια κλπ από την μια μεριά, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και τους δωρητές ε, ιδιωτικού τομέα. Τελικά, για πέστε μας. Ποιο ε, διαμορφώνει περισσότερο τις ε, πολιτικές και τις προτεραιότητε, Και άπαξε και κάποιος από αυτούς ενεργεί στα πλαίσια προτεραιοτήτων μας, ε, από ποια κατηγορία κυρίως γίνεται αυτό. Α, ο κύριος Πόγκα έχει άλλη μια ερώτηση. Δεν πρόκειται περί ερωτήσεως, Πρόεδρε. Απλώς μία σκέψη μου. Επίσης να ευχαριστήσω και τους δύο προσκεκλημένους μας. Ήταν την ενημέρωση που μας προσέφεραν. Ξέρετε, είμαι ο εισηγητής και σας τονίζω ότι συμφωνώ ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τρεις αρρώστιες που σκοτώνουν όπως είπατε και τις οποίες δεν υπάρχουν εμβόλια. Συμφωνώ ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα στο μέτωπο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Παμίλου Πρόεδρος. Κύριε Σβένσον, έχετε εσείς το λόγο. Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ αξιόλογες αυτές οι οι ε, Πάρε μιλάγατε γρήγορα, δεν ξέρω, ίσως ε, έχω γεράσει. Τέλος πάντων, θα ζητήσω ότι τέλο. τέλος, όταν τελειώσει η συνεδρίαση. Και θα σα πω για ένα μεγάλο πλεονέκτημα, το ότι μπορούμε να επικοινωνούμε με αποτελεσματικό τρόπο. Έχουμε τώρα τα στοιχεία για το πόσοι έχουν εμβολιαστεί Δεν σκέφτω πάντα στα όσα κάνουμε για την αυτοσιακή βοήθεια. Το θέμα είναι όμως, ξέρετε όλη μου τη ζωή έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό και όταν διαβάζω κείμενα σαν και αυτό νιώθω ενθάρρυνση. Τώρα, μπορεί να υπάρξει έτσι σωστή ενημέρωση η οποία επιδέχεται βελτίωση. Αλλά αν κατάλαβα καλά τα στατιστικά στοιχεία, νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες χώρες να εμπλακούν. Εσείς το καταφέρετε αυτό. Θέλετε 14 χώρες να πάτε στις 33. Πολύ μεγάλο άλμα. Δεν ξέρω αν θα αποδώσει. Αλλά πάντως αν το καταφέρετε τότε αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι περισσότεροι να συνειδητοποιήσουν σε ποιο σημείο βρισκόμαστε γιατί έχουμε ήδη κάνει μια μακρά πορεία. Κόρτες Λάστα. ευχαριστώ και συγχαρητήρια για το τρόπο που έχετε επιτελέσει. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Εδώ και χρόνια ε, αντιμετωπίσαμε το ζήτημα του AIDS Είχαν τότε είχαν 15.000 δολάρια, χρειαζόταν η, ε, ε, η, η, θεραπεία, τώρα ε, χρειάζονται 20-30 ευρώ και νόσημα για να εξυπηρετηθεί τόσο κόσμο, όλο τον κόσμο. Άρα μακάρι όλο δυο τη αρρώστια να τα πράγματα να είναι η αντιμετώπιση πιο γαλήνια, πιο αποτελεσματική. Είπατε λοιπόν εσεί, για το χαμηλό κόστο, των σχετικών φαρμάρων για του οποίου. είπατε. Για πετε μα τι γίνεται, δουλεύετε με γενώσιμα γιατί Ξέρουμε όλοι τι γίνεται με την ε, έρευνα. Συνήθως το κράτος και τα πανεπιστήμια εμπλέκονται σε τέτοιες επενδύσεις. Συνεργάζεστε με βιομηχανίε. Πώς καταφέρετε να βρίσκετε φάρμακα σε τόσο και τιμέ, Η πρώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει να θέσει κάποια ερώτηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι τώρα, ίσως αργότερα θα κάνω κάποια σχόλια. Ευχαριστώ πολύ όμως. Εντάξει, θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας. Δεν ξέρω ποιος θέλει να λάβει το λόγο πρώτος. Κύριο Μπέρκλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ερωτήματα που έχετε θέσει. Για το πρώτο ερώτημα. <clears throat> τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι σημαντικά για τα εμβόλια όπως είναι για τα φαρμακευτικά συσκευάσματα. Πολλά εμβόλια, ε, για τα εμβόλια το σημαντικό είναι η τεχνογνωσία γιατί είναι τόσο δύσκολο να φτιάξει κανείς ένα κέντρο εμβολιασμού, ένα, μια παραγωγή εμβολιασμού, ένα φάρμακο είναι κάτι το οποίο μπορεί να φτιάξει κανείς εύκολα, αλλά το εμβόλιο είναι ζωντανό. Είναι μια ζωντανή ουσία, γι' αυτό είναι πολύ λίγοι οι κατασκευαστές των εμβολίων. Γι' αυτό το κόστος της ανάπτυξης τεχνογνωσίας είναι το πιο σημαντικό. Για την περίπτωση της υπατήτηδος γ, παραγωγής χάρη οι εταιρείε που είχαν κάποιο, κάποια ευρεσιτεχνία δεν τη δίνανε σε άλλου και αυτό σημαίνει ότι οι μικρότερε εταιρείε δεν μπορούσαν να κάνουν έρευνα και αυτό εμπόδισε την πρόθεση τη επιστήμη. Σε μερικέ περιπτώσει λοιπόν η πνευματική διοκτησία είναι ένα εμπόδιο αλλά όχι πάντα. Το δεύτερο ερώτημά σα για του ιδιωτικού θεωρητέ. Έχουμε ενδιαφέρουσα ε, μορφή διοικητικού συμβουλίου και το Ίδρυμα Gates, Bill Gates έχει εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και η Κομισιόν και αναπτυσσόμενες χώρες, κοινωνία των πολιτών και φαρμακευτικέ εταιρείε και από το βορρά και από το νότο. Η ιδέα μα είναι να είναι όλοι εμπλεκόμενοι στο διοικητικό συμβουλίο μα. Επομένω, ένα ίδρυμα όπω το ίδρυμα Gates δίνει μεγάλη χρηματοδότηση <clears throat> χρηματοδοτεί κυρίως την κέρια λειτουργία του οργανισμού και τα σημεία τα οποία έχουν συμφωνηθεί από όλους. Και επομένω, έχει μεγάλη επιρροή ως δωρητής, αλλά δεν ελέγχει τη δράση του οργανισμού μας και δεν μπορεί να αλλάξει την ατζέντα μας. Ο συνάδελφός μου θα μιλήσει για το EDCTP. Απλώς ήθελα να πω ότι εγώ ήμουν επικεφαλής του οργανισμού που είχε να κάνει με τα ε, εμβόλια για το AIDS και είναι πολύ σημαντικό για μας να υπάρξει ανάπτυξη στα θέματα αυτά σε επίπεδο ερευνητικό και πανεπιστημιακό και μετά φυσικά έρχονται στον κάβι που μπορεί να τα διανύμει στον πληθυσμό. Για το ερώτημά σας, για την διάδοση των πληροφοριών. Αυτό είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική προτεραιότητα. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί είναι μετρήσιμο και ποσοτικοποιήσιμο το έργο μας και δεν μπορεί να επηρεαστεί από τη διαφθορά. Άλλοι τομείς ανάπτυξης που είναι πολύ σημαντικοί, ε, όπως είναι η ευκυβερνησία, είναι πολύ πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η ευκυβερνησία. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι οι ίδιες οι χώρες, οι εμπλεκόμενες να δώσουν προτεραιότητα στα θέματα αυτά μέσω των Υπουργείων Οικονομικών για να δούνε ποιο πρέπει να είναι το κόστος των παρεμβάσεων και ποιες οι προτεραιότητες. Χρειάζεται λοιπόν μια συνολική κίνηση σε όλες τις χώρες μας, γιατί ακόμα και στις χώρες μας υπάρχουν πολλές φορές προβλήματα με τα εμβόλια και είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε αυτές τις παρεμβάσεις που σώζουν ανθρώπινες δομές, ζωές. Η Σουηδία συγκάλεσε μια συνδιάσκεψη πριν από δύο εβδομάδες για τα θέματα αυτά. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τις πληροφορίες, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Για τα γενώσιμα τέλος. Δεν υπάρχουν γενώσιμα εμβόλια, υπάρχουν γενώσιμα φάρμακα, αλλά με το να δημιουργήσουμε μια αλλαγή νοοτροπίας, να δημιουργήσουμε μια αγορά για τα προϊόντα αυτά, έχουμε πλέον βιομήχανους από τις χώρες, τις που μπαίνουν στην αγορά, οπότε τον Γκάβι έχει προμηθευτές από στην αρχή είχε τέσσερις από τον αναπτυγμένο κόσμο και ένα από υποανάπτυξη χώρες και τώρα έχουμε 13 κυρίως από αναπτυσσόμενες χώρες, Σενεγάλη, η Ινδία, ε, Ινδονησία, η Κίνα έχει μπει στο παιχνίδι. Όλα αυτά δημιουργούν ένα θετικό ανταγωνισμό και αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν οι τιμές αλλά θα υπάρχει καλή αγορά για τα εμβόλια. Αυτό θέλουμε λοιπόν να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να επαναλάβω ότι όταν η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδασε το έργο του Γκάβη, η κυβέρνηση βρήκε ότι ήταν πάρα πολύ καλό το έργο της Γκάβη και αξίζει τα χρήματα που παίρνει. Μια ερώτηση αφορούσε το πώς ε, τα ιδρύματα και οι δωρητές του ιδιωτικού τομέα συμμετέχουν χωρίς να προσανατολίσουν τις δραστηριότητες εκεί που θέλουν. Όπως είπε και ο κύριος Μπάκλη, ε, το σημαντικό είναι η διακυβέρνηση και η διασφάλιση ότι τα ιδρύματα ή οι δωρητές του ιδιωτικού τομέα συνεργάζονται μέσα στο πλαίσιο που έχει θεσπιστεί πολυμερός. Κάποια παραδείγματα. Στην ε, Λονουσία έχουμε το εμβόλιο ε, TSS που αναπτύχθηκε στο Βέλγιο από την GSK και στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και στην Αφρική. Η GSK εργάζεται μέσα σε ένα πλαίσιο, όχι μόνη της, ε, ανεξάρτητα. Επίσης, ανέφερα κάποια πολύ φθηνά φάρμακα για τροπικές νόσους. Ε, και στο πίσω μέρος της έκθεσης ε, ε, υπάρχει κατάλογος όλων των φαρμακευτικών εταιριών και των δωρεών της τελευταίας δεκαετίας που ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δισκία. Τα φάρμακα είναι φθηνά, αλλά χωρίς τις δωρεές στα προγράμματα, γιατί αυτά οι δωρές γίνονται βάσει προγράμματος και για κάποιο συγκεκριμένο ε, πρόγραμμα. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να καταπολεμήσουμε τις τροπικές νόσους. Ε, αυτό που, είπαμε για τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικό. Ε, τα δεδομένα για την λονοσία είναι αμφισβητούμενα. Πιστεύουμε ότι ο αριθμό των θυμάτων μειώθηκε από ένα εκατομμύριο το χρόνο πριν από μία δεκαετία στο, στους 660.000. Άλλοι τα αμφισβητούν, δεν ξέρουν και για, ε, για μια νόσο όπως η ελονοσία που παρουσιάζεται με πυρετό σε επιτοπλίστονο σύμπτωμα, όταν βλέπουν κάποιοι παιδί με πυρετό θεωρούν ότι έχει ελονοσία, να μπορεί να έχει πνευμονία ή κάποια άλλη εμπειρετή νόσο, αλλά το παρουσιάζουν ως και το ταξινομούν ως ελονοσία. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε καλύτερα τη, περισσότερο συλλογή δεδομένων, ούτω ώστε να στοχεύσουμε τις παρεμβάσεις μας ε, καλύτερα και να έχουμε καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους. Ε, είπατε ότι πρέπει να συμμετέχουν περισσότερες χώρες. Συμφωνώ όσο δεν πάει. Ε, μάλιστα δεν ήθελα να ε, είμαι επιθετικός στην έκθεση για την ελονοσία που τη λέμε το Σταυροδρόμι. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχει μεγάλη πρόκληση και υπάρχει κίνδυνος να υπαναχωρήσουμε ε, και να κάνουμε βήματα προς τα πίσω στη ε, μάχη μας κατά της ελονοσίας. Θέλω λοιπόν να ε, κρούσω κόδωνα κινδύνου προς τη διεθνή κοινότητα γιατί χρειαζόμαστε διπλάσια κονδύλια από ό,τι θα έχουμε για να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά την ελονοσία. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα και χαιρετίζω την πρόταση που έγινε και πάνω στην οποία εργάζεται ο κ. Σπόγκα. Τέλος, ο ρόλος των πανεπιστημίων και της έρευνας. Ε, πάρα πολύ σημαντικός, όπως καταλαβαίνετε. Ε, για παράδειγμα, στις παραμελημένες τροπικές νόσους στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε και στο Λίβερπουλ και στο Λονδίνο και το Imperial College στο Λονδίνο όλοι αυτοί συνεργάζονται στο θέμα των παραμελημένων τροπικών νόσων για να αυξήσουν την ικανότητά μας στις ενδυμικές χώρες όπου χρειάζεται περισσότερη έρευνα στις χώρες όπου είναι ενδυμικές οι νόσοι αυτές γιατί έχουμε πολύ λίγες δυνατότητες ε, σήμερα αν ας πούμε έχουμε τη ε, φιλορίαση των λεμφαδένων ε, υπάρχουν πολλοί ε, λίγοι ειδικοί σε αυτή την όσο Χρειάζεται λοιπόν εκπαίδευση, κατάρτιση και είδατε στο πρόγραμμα δίνεται μεγάλη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και για την αύξηση των ικανοτήτων που διαθέτουμε που είναι πολύ ζωτικό θέμα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λουβρό, κύριε Βέκλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψή σας στην Επιτροπή Αναπτύξεως σήμερα. Καλή συνέχεια όσον αφορά το έργο σας, όσον αφορά την προσπάθειά σας κατά αυτών των ασθενειών. Αφορά και τις τρεις επιτροπές και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Donc, euh, nous avons des documents que vous pouvez prendre à la, à la sortie tout à l'heure. Nous allons continuer notre réunion. Euh, το επόμενο σημείο της ε, έχει να κάνει με το προηγούμενο θέμα, δηλαδή αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης σαν δεύτερο πρόγραμμα, και σχέσεις των ευρωπαϊκών χωρών και ε, την ανάπτυξη, την, την, ε, για τα κλινικά πειράματα τις κλινικές δοκιμές. Είμαστε αρμόδια επιτροπή μαζί με την Ήτρα. Ο κύριος Πόγκα είναι ο ε, συντάκτης και έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας παρουσιάσω με λίγα λόγια αυτή την γνωμοδότηση που συνέταξα για το καινούργιο πρόγραμμα όσον αφορά αυτές τις δοκιμές. Εδώ ξεκινούμε μια εταιρική σχέση μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και αναπτυσσομένων χωρών όσον αφορά αυτές τις δοκιμές, τις κλινικές. Επόκειται για κάποιες ε, μολυσματικές ασθένειες και το 2003 ξεκίνησε αυτή η εταιρική σχέση για πρώτη φορά. Το NDSNDP ήταν το πρώτο πρόγραμμα και είχαν συμμετασχεί 14 χώρες με Νορβηγία, η Ελβετία και 48 χώρες ε, της Αφρικής τη Σαχάρας και λόγω αυτού του προγράμματος στην ΕΣΕΠΕΜΠΕ 1 είχαμε κάποιες ε, καινούργιες ε, μορφές για τις κάλυψεις και είχαμε και επίσης και κατάρτιση και εκπαίδευση 400 περίπου Αφρικανών ιατρών. Πάρα πολύ θετικό θεωρώ το ότι τώρα θα ε, δοθεί παράταση σε αυτό το πρόγραμμα δοθεί ένα δεύτερο τέτοιο πρόγραμμα, θα καλύψει μια δεκαετία και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες ε, ιατρικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με τις χώρες αυτής της, ε, αυτού του τμήματος της Αφρικής, συντονισμός των εθνικών προσπαθειών και επίσης θα συνεργαστούν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα δωρητές του δημοσίου και δυτικού δικαίου. Επίσης έχουμε τους του Γκάβη και έχουμε τον πρόεδρο ε, που, που μας μίλησε προηγουμένως όσον αφορά την λονοσία και τις ε, παραμελημένες ασθένειες οπότε θα πρέπει επομένως να συνεχίσουμε τις επενδύσεις μας στην έρευνα να μπορέσουμε να ξεύρουμε και να επινοήσουμε καινούργια φάρμακα ε, το AIDS, η ελονοσία οι φηματίε σκοτώνουν πάνω 5 εκατομμύρια χρόνια, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε σταυρώνουν τα χέρια. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση αυτών των ε, για αυτέ τι ασθένειε. Έχουμε εδώ πέρα ένα σωρό τροπολογίε και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε ένα κείμενο πιο συνεκτικό ε, και να υπάρχει συνέπεια μεταξύ παραρτημάτων και κυρίω σώματο όσον αφορά κάποιε αρρώστιε ε, από αυτέ, όπω το AIDS, τη φυματίωση και κυρίως να στην προσοχή μας όσον αφορά τις ασθένειες που έχουν κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Πάντως θα πρέπει να, είμαστε, να καταβάλουμε κάμετες προσπάθειες για την έρευνα για τις ασθένειες αυτές που πλήσουν τους πιο ευάλωτες της κοινωνίας. Επίσης θεωρώ θετικό το ότι η Επιτροπή στην πρότασή της αυξάνει σημαντικά την οικονομική συμβολή της ε, Ένωσης. Μιλούμε για 200 εκατομμύρια το 2003 και τώρα για το έντεσε τεπέ υπαρθμόν 2 θα έχουμε 683 ε, εκατομμύρια. Πάρα πολύ καλό μήνυμα αυτό το ότι δηλαδή η Ευρώπη ανεβάζει τον, τον, τον πύχη, προσπαθεί περισσότερο να βοηθήσει τις χώρες νοτιού της αγοράς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ουσιαστική συμβολή της ε, Επιτροπής θα πρέπει να καταργήσουμε αυτά τα κατόφλια του άρθρου 2 παραγράφου υπαριθμών 1. Εκεί που λέμε για το πώς θα δημορφωθεί η συμμετοχή, αυτό εδώ πέρα δεν είναι δόκιμο γιατί έτσι θα μειωθεί ε, η δυνατότητα κάλυψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όλου του προβλημένου ποσού των 683 εκατομμυρίων. Επίσης, λέω σε, πολλά, σε πολλές τροπολογίες θα πρέπει να είμαστε συνεπείς με τους στόχους της ανάπτυξης. Επίσης θα πρέπει όσον αφορά αυτές τις δράσεις να κάνουμε αυτά τα οποία ήδη έχουμε εξαγγείλει στο πλαίσιο του προγράμματος και όλοι να κινητοποιηθούν όσον αφορά αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών. Επίση, διευκρινίζω ότι η έρευνα θα πρέπει να καλύψει τι ανάγκε των οψημένων χωρών, αλλά επίση και την υποχρέωση ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κάποιος τρόπο ιατρική αντιμετωπίσεω. Και ακριβώ αυτέ οι έρευνε των των χωρών θα πρέπει να ανταποκρίνονται όσο γίνεται καλύτερα στι ανάγκε των αντισωμένων χωρών και ιδίω νοτιού Σαχάρα. Και θα πρέπει επίση να εμβαθύνουμε στο θέμα τη διακυβέρνηση για το νέο πρόγραμμα ΕΝΤΕΣΕΠΕΤΕ 2. Στο τρίτο παράδειγμα αναφέρονται κάποιες σχέδια με την διακυβέρνηση όσον αφορά την αρχιτεκτονική αυτού του νέου προγράμματος. Λέει για μια συνέλευση, γενική συνέλευση, διοικητικό συμβούλιο και γραμματεία, όμως τίποτα δεν λέει όσον αφορά την σύνθεση αυτών των οργάνων, ούτε τους τρόπους λήψης των αποφάσεων. Οπότε μου λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το, το πρόγραμμα NDSTP2 πρόκειται να αναδεχθεί την δομή, την νομική που προβλέπει το Ολλανδικό δίκαιο. Γι' αυτό δεν λέγεται τίποτε άλλο. Πάντως θα πρέπει αυτό να διευκρινιστεί. Πώς θα γίνεται η διακυβέρνηση σχετικά με αυτό το πρόγραμμα. Περιμένω πώς και πώς να μου τα διευκρινίσει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τι θα γίνει στο μέλλον. Για κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες δεν συνάδουν προς το τρίτο παράδειγμα. Και μιλώ κυρίως για το δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, εκεί δηλαδή που ακόμα και που, ε, και, εκεί που έχουμε την, την απαρίθμηση των στόχων. Τρίτη, 3 Δωδεκάτου το μεσημέρι, νέοι προθεσμοί για τις τροπολογίες. Κύριε Πόγκα, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Κύριε Φιονόρε, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ ιδιαίτερα τον κύριο Πόγκα για την έκθεσή του. Εγώ είμαι και στην Επιτροπή ΔΕΒΕ και ΙΤΡΕ Σχεδόν εισηγείται για τα θέματα αυτά. Τα εμβόλια είναι πολύ αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με τον κόστο για να αποτρέψουν θανάτους χωρίς λόγο και ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο εκατομμύρια παιδιά που πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειε που μπορούσαν να προληφθούν από τα εμβόλια. Η υποσαχάρη Αφρική είναι αυτή η οποία πλήττεται περισσότερο από ασθένειε όπω η φυματίωση, η ελονοσία, το AIDS κτλ. και άλλε ακόμα πιο άγνωστες και παραμελημένε ασθένειε. Ξέρουμε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείε γενικά έχουν ε, δισταγμού όταν κύρια αγορά του είναι αναπτυσσόμενε χώρες γιατί εκεί δεν έχουν τόσο υψηλά κέρδη. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να μπορέσουμε να δώσουμε τα εμβόλια μέσα από το EDCTP σε όλες αυτές τις χώρες και να εξασφαλίσουμε ότι είναι προσιτά για τους πληθυσμούς που τα χρειάζονται περισσότερα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Πόγκα για τις τροπολογίες που έχει καταθέσει και θα καταθέσω και εγώ βέβαια μερικές θα πρέπει να δούμε πώς το EDC TP2 μπορεί να προχωρήσει περισσότερο και να βασιστεί στις επιτυχίες του EDC TP1. Κάτι λοιπόν το οποίο είναι πολύ σημαντικό για όλους μας είναι να καλύψουμε περισσότερες ασθένειες πέραν του αυτό που καλύπτονται στο πρώτο EDC TP. Είχα τη μεγάλη χαρά να μπορέσω την προηγούμενη εβδομάδα στην ε, συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στην αντίσαβεβα να πάω σε ένα νοσοκομείο και γνώρισα τον καθηγητή Άσρατ που είναι ε, ειδικό στην δυσμανίαση και μου εξήγησε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο πληθυσμό. Είναι μια τρομερή ασθένεια που είναι πολύ διαδεδομένη στο χώρο της υπαίθρου και κατά 98% είναι θανατηφόρα ασθένεια. Είναι κυρίως τα παιδιά λοιπόν που πλήττονται από αυτήν. Η μόνη <clears throat> θεραπεία που έχουν αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ τοξικού χαρακτήρα. Σημαίνει ότι πρέπει να μείνει κανείς στο νοσοκομείο και με ε, ενέσεις να δώσουν αυτό το φάρμακο και να παρακολουθούν τον ασθενή γιατί είναι πάρα πολύ τοξικό το φάρμακο. Δεν υπάρχει καμιά άλλη θεραπεία. Λείπουν λοιπόν στοιχεία ακόμα και σε επίπεδο βασικό ερευνητικό για να ξέρουμε πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε καλύτερα προτού αντιμετωπίσουμε αυτές τις ασθένειες. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή να συναντήσω αυτόν τον ιατρό που μου τόνισε πόσο σημαντικό είναι το έργο μας για όλα αυτά τα θέματα. Το σημαντικό εδώ είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα κρατήσουμε αυτά τα 183 εκατομμύρια ευρώ που έχουν προσδιοριστεί για αυτό το πρόγραμμα και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα ήταν εσφάλμα να έχουμε μια τεχνητή κατανομή μεταξύ συμμετεχών των ίδιων κρατών μελών και νέων κρατών μελών, γιατί αυτό που θα συμμετέχουν, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη δαπάνηση ορισμένων ποσών. Τώρα βλέπω κάποιους ε, αριθμητικούς στόχους που μου φαίνονται κάπως αυθαίρετοι. Πρέπει εμείς να δώσουμε την έμφαση στην ε, ποιότητα και στο προσιτό των θεραπείων και όχι απλώς να κάνουμε ε, προσπάθειες να πιάσουμε κόσμιους αριθμητικούς στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Στυρολιέν. Χωρίς μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα εξακολουθούν να πεθαίνουν εκατομμύρια ανθρώπων, κυρίως παιδιά, από ασθένειες που οφείλονται στην ε, ένδια μεταξύ των οποίων και η ελληνοσία. Η υποσαχάρη Αφρική πλήττεται ιδιαίτερα από αυτές τις ασθένειες. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των ατόμων που πλήττονται από τα έτσι στην υποσαχάρη Αφρική, τα δύο τρίτα περίπου. Από την άλλη πλευρά υπάρχει έλλειψη φαρμάκων και αναποτελεσματικότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρώτος ε, παγκόσμιο εταίρος στον τομέα της ε, υγείας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της περίθαλψης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με την ανανέωση του προγράμματος εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτυσσομένων χωρών για τις κλινικές δοκιμασίες, για το οποίο συζητούμε σήμερα, έχει μια μεγάλη σημασία. Το πρώτο πρόγραμμα, το EDCTP, e ήδη κατήγαγε σημαντικά αποτελέσματα, υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις στις ιατρικές θεραπείες, ιδίως για να αντιμετωπιστεί το hiv Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν το έργο αυτό και να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το έργο του και νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να διευρύνουμε περισσότερο το εύρος εφαρμογής των προσπαθειών μας και να υπάρξει μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων αναπτυξιακών φορέων και χαιρετώ τι διευκρινήσει σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και αυτό το οποίο λέει ο εισηγητής μας, δεν πρέπει να μιλάμε για χορηγούς, αλλά για εταίρου, Εκεί προτιμώ τη διατύπωση της Κομισιόν και θα ήθελα να υπάρξει και μια διεύρυνση του αριθμού των ασθενειών που καλύπτουν το πρόγραμμα, ιδίω σε αυτέ οι οποίε πλήττουν ιδιαίτερα τα παιδιά και θέλω να τονίσω την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη ε, σχέση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό της ανάπτυξης ώστε αυτά τα οποία δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα παγκόσμια ταμεία για την αντιμετώπιση των αστεών να δίνουν ιδιαίτερα έμφαση στην μεγαλύτερη χρηματοδότηση της έρευνας προς όφελος των πληθυσμών στις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτές τις ασθένειες. Και επίσης το νομικό εργαλείο η νομική μορφή για τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων δεν έχει ακόμα καθοριστεί από την έκθεση και αναπόκειται από, στην Κομισιόν να διευκρινίσει το σημείο αυτό για να μην υπάρχουν προβλήματα στα μελλοντικά προγράμματα. Ευχαριστώ. Monsieur. Ευχαριστώ κύριε Τυροντιάν. Ο επόμενος ομιλητής, ναι, ναι, α, συγγνώμη, από την Επιτροπή, αλλά δεν είμαι στην ΤΕΒΚΟ, είναι η... Είμαι από μια άλλη γενική διεύθυνση, από την ε, Γενική Διεύθυνση για την Έρευνα στον τομέα αυτό. Η Κομισιόν θέλει ευχαριστήσει τον κύριο Πόγκα για την ε, έκθεσή του που υποστηρίζει την πρόταση της Κομισιόν για το EDCTP. Όπως ξέρετε το EDCTP 2 είναι μια αναβαρχίδα για την Κομισιόν, μια εμβληματική πρωτοβουλία με τον ορίζοντα 2020 και ιδιαίτερα είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές προκλήσεις σε κοινωνικό επίπεδο με το να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με τις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής για να υπάρχει και μεγαλύτερη πρόοδο στην υγειονομική περίθαλψη. Η έκθεση και οι τροπολογίες της είναι μια σημαντική συμβολή στη διαθεσμική ανταλλαγή απόψεων και η Κομισιόν χαιρετίζει ιδιαίτερα την θέση του εισηγητή, ο οποίος θέλει να δώσει μεγαλύτερη σημασία στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια δράση υπέρ της υγείας, όπως ελέγχθηκε από τους ε, Βουλευτές, το 1 τέταρτο των συνολικών επενδύσεων στην παγκόσμια υγεία γίνεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Επίση όμω είναι σημαντικό να προωθήσουμε τι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει και μεγαλύτερη ορατότητα και ιδίω ορατότητα του EDCTP όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην υποσαχάρια Αφρική και παντού. Η Κομισιόν κατανοεί ότι η δράση του EDCTP θα πρέπει να ανταποκρίνεται στι ανάγκε των αναπτυσσομένων χωρών αλλά και στι δεσμεύσει Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την παγκόσμια υγεία και το οποίο να είναι συμπληρωματικό με τι υπόλοιπε ενέργειε συνεργασία για την ανάπτυξη που ε, ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τονίσουμε ιδιαίτερα ότι πρέπει να υποστηριχθούν οι ιατρικές δράσεις στο EDC-TP, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι προσιτές οικονομικά, ασφαλείς και αποδοτικές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο προτείναμε ένα διευρυμένο προϋπολογισμό για τα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα το καταστατικό της μελλοντικής αυτής τελικής σχέσης, της ε, σχέση αυτής, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί μεταξύ των συμμετεχών των κρατών. Η Κομισιόν έχει υποδείξει ορισμένες ε, <clears throat> αναντιστοιχίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ των απόψεων των διαφορών πλευρών. Ξέρετε ότι και τα κράτη-μέλη έχουν ζητήσει τουλάχιστον μία αλλαγή για το παράτημα 3. Επομένως παρακολουθούμε από κοντά όλα τα θέματα αυτά για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη συνεκτικότητα μεταξύ του καταστατικού και των δράσεων και αναμένουμε την απόφαση για το παράρτημα 3 εν καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάω και πάλι στον εισηγητή. Αν θέλετε κύριε Πόγκα να κλείσετε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μην με θέλω να ευχαριστήσω του που έλαβαν λόγο και τον κύριο Τυρολίνη και τους άλλους για, σε σχέση με τις τροπολογίες όπως είπαμε αύριο εκπνέει η προθεσμία 3 Δεκεμβρίου ευχαριστώ Η πρόεδρος ευχαριστούμε κύριε Πόγκα πρέπει να συζητήσουμε α μάλιστα σας υπενθυμίζω το είπε ήδη ο κύριος Πόγκα ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για αυτή την έκθεση εκπνέει αύριο 3 12 την Μεσημβρίου. Μάλιστα και το επόμενο θέμα ε, είναι λίγο προβληματικό διότι ο κύριος Ζαχαραντήλ ακόμη δεν έχει... Α, εδώ είναι. Α, ήρθε. Να, τόσο. Ωραία. Οπότε. Να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις τροπολογίες όσον αφορά την έκθεση της ε, ΑΦΕΤΟΥΝΙΑ που είναι η κυρίως Επιτροπή όσον αφορά τον ρόλο του Πακιστάν και τις ε, σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Θα γίνει η ψηφορία σήμερα κιόλας, ε, αλλά θα πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Ζαχράντιλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. θα είμαι απλός και σύντομος για να καταλήξουμε σε συμφωνία σε όλες τις περιπτώσεις για τις τροπολογίες. Εμείς τις δεχτήκαμε σχεδόν όλες με τρεις εξαιρέσεις. Ετοιμάσαμε και μια συμβιβαστική τροπολογία. Οπότε μόνο την 11 και τη 12 προτείνω να μην τη δεχτούμε. Όχι τόσο λόγω του περιεχομένου, αλλά λόγω των συμφραζομένων νομίζω ότι δεν αντικατοπτρίζουν το θέμα και προτείνω να καταψηφίσω με τη 17. Κατά τα άλλα είμαι ευτυχής από τις τροπολογίες όλων των συναδέλφων και τους ευχαριστώ για τη φιλική ατμόσφαιρα που επικράτησε νομίζω ότι συνέβαλαν πολύ επικοδομητικά στην τελική μορφή του κειμένου. Ευχαριστώ. Καταψηφίζουμε 17, αποχή στην 11 και 12 λοιπόν. Ευχαριστώ. Επιθυμεί κάποιος το λόγο, έχετε ερωτήσεις. Όχι από ό,τι φαίνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μήπως Όχι. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε πριν την προηγούμενη ώρα. Δεν προβλέπεται. Οπότε θα διαγώσουμε μέχρι τις 5.30. Θα πούμε σε λίγο. Έλα ματούλα. Ach. Βγάλτε τις κάρτες σας παρακαλώ για να ψηφίσετε. Όχι τις πιστοτικές ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Ναι, ευχαριστώ. Σε ένα λεπτό ξεκινάμε. 17 h 5.30 είναι, οπότε θα προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Βιαζόμαστε ορισμένοι από εμά. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε τη δοκιμαστική ψηφοφορία. Κάποιος λείπει εδώ. Κάποιος δεν έχει ψηφίσει. Γκέρενς. Ναι. Όχι. Ναι, ναι, απλώς, απλώς δοκιμαστικό ήταν αυτό. Ήταν δοκιμαστικό κύριε Γκέρνς. <laughs> ναι, ναι, όχι δεν λέω τίποτα για τα χαρτιά. Ξεκινάμε με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την πορνεία και τις, και τις συνέπειες για την ε, ισότητα εδώ και γυναικών. Παράγραφος τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίζεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 3. Υπέρ κατά αποχές από 4 υπέρ όλες μαζί από τις 4 έως τις 10 ναι όλοι υπέρ κατά αποχές όλες μαζί εγκρίνονται τελική ψηφοφορία ηλεκτρικά ναι υπέρ κατά και τώρα ηλεκτρονικά άρχεται πέρας εγκρίνονται. Ευχαριστώ. Περνάμε στην ψηφοφορία για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο από τη βάση της συμφωνίας της 5 Νοεμβρίου. Εδώ χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Ψηφίζουμε λοιπόν για την έναρξη των διαπραγματεύσεων υπέρ κατά αποχές δεκτή ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Αυτή είναι η διαδικασία, όπως μου είπαν οι συντονιστές. Πέρασε. Ψηφίζουμε λοιπόν για τη σύνθεση της ομάδας διαπραγμάτευσης. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι ανόητο να ψηφίζουμε δύο αλλά έτσι είναι η διαδικασία. Πέρας. Τέλεια, εγκρίνονται. Ωραία. Έχουμε τώρα την έκθεση του κυρίου Ζαχραντέλ για τον Πακιστάν και τον περιφερειακό του ρόλο. Ναι, παρακαλώ. Μπορούμε να ψηφίσουμε την 1 ως τη 10 από κοινού, όλες μαζί. Συλλήβδιν, βεβαίως. Από 1 ως την 6. 1 ως την 6. Ναι, άφησα να τελειώσω. Λοιπόν, 1 με 6. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 7. Όχι, οι 7 και οι 8 εκπίπτουν. Ναι, ναι. Α, ήταν κρυφά αυτά. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. 10. Υπέρ κατά αποχές δεκτή, 11 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά, 11. Πέρας. Εγκρίνεται. ναι, δεν σηκώσατε τα χέρια σε εγκαίρος. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. 17. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία λοιπόν. Με ανατασχυρών υπέρ, ε, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας. Ο κύριος Μπέρμαν καθυστέρησε. Κύριε Γκέρνς, θέλετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε. Συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι ανόητο να ψηφίζουμε δύο φορές. Θα ήθελα να σας ζητήσω να υπάρξει κάποια τροποποίηση αυτής της διαδικασίας. Δεν σημαίνει ότι επειδή το κάνουμε στο παρελθόν εξακολουθεί να είναι ευφυές να το κάνουμε και στο μέλλον. Μου λένε ότι αυτό ήταν μια απόφαση των συντονιστών των Φρασίνων και της ε, Άλντε, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει μια άλλη η οποία είναι κάπως παράδοξη για να το πω ε, ευγενικά. Μπορούμε να επανέλθουμε λοιπόν. Donc les votes sont terminés. Mais... Τέλειωσαν οι ψηφοφορίε, αλλά δεν μπορείτε να φύγετε. βρισκόμαστε τώρα. Σας παρακαλώ, για καθίστε. Δεν έχουμε τελειώσει. Περνάμε στην ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο γνωμοδότησης για ένα μη νομοθετικό μια μη νομοθετική πρωτοβουλία της ε, Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για τις επιστροφές και την εφαρμογή της οδηγίας για τις επιστροφές. Κύριε Μπέρμαν, μιλάτε πολύ δυνατά, δεν σας ακούει κανένας. Η κυρία Σύμπερια Στράμ δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρούσα για να παρουσιάσει το σχέδιο. Ο κύριος ε, Μη... Ο κύριος Κάσμα καθιστά λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Σίμπερ και Άστον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να σας πω ότι η Μπίργκετ ζητεί να την συμπαθήσετε γιατί είχε μια υποχρέωση πάρα πολύ σημαντική στην εκλογή της περιφέρεια. Οπότε και εγώ θα προσπαθήσω να την ε, αντικαταστήσω και να σας παρουσιάσω αυτό το σχέδιο κειμένου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα γιατί έχουμε την προβληματική που έχει αναπτυχθεί για την πολιτική της μετανάστευσης και θα πρέπει να δούμε τι έγινε πριν από λίγες εβδομάδες ή στην Λαμπεντούζα. Ε, αυτοί όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν είναι κρίσιμη κατάσταση. Πολλές φορές γίνεται κατάσταση και τραγική νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε πόσο σημαντική υπόθεση είναι η στην λαμπεντουζα αυτοι ολοι οι ανθρωποι οι οποιοι φευγουν ειναι κρισιμη κατασταση Πολλέ φορες γινεται κατασταση και τραγικη νομιζω οτι ολοι καταλαβαινετε ποσο σημαντικη υποθεση ειναι Η κυρία Σνίμπερ έχει τρεις άξονες στο κείμενό της. Πρώτα πρώτα η σημασία της υποβοηθούμενης εκούσιας επιστροφής. δηλαδή να δει πώς θα έχουμε μεγιστοποίηση της ποιότητας και όχι επικέντρωση, εστίαση της προσοχής ή στην ποσότητα, γιατί θα πρέπει να γίνεται επιστροφή με τρόπο ανθρωπιστικό και θα πρέπει να τη τηρούνται, αν είναι το σεβαστό των ανθρώπινων στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να κάτσουμε και να ξανασκεφτούμε τι θα πει χώρα ε, τέρος, ε, τι θα πει η χώρα προέλευση ποιε είναι προτεραιότητε, τι γίνεται με τι τοπικέ αρχέ. Ε, και όσον αφορά τα ανθρώπινα είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά τα προβλήματα τη εκούσια επιστροφή και επίση για την επανεισδοχή. Αυτές οι συμφωνίες ε, είναι το δεύτερο σημείο που σχέση με η έκθεση και επίση όσον αφορά το νομικό Καθεστώ, η κυρία Σνίμπερ λέει ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο εκτέλεσης εφαρμογής του πρωτοκόλλου, πολύ σημαντικό αυτό, και τελευταίο όλα σημαντικό. Η... Συντάξασα την έκθεση, Τονίζεται στις πτυχές της ε, ανάπτυξης, σημαντικό για την Επιτροπή μας, έχει απόλυτη άποψη ότι καμία πολιτική μετανάστευση δεν θα πρέπει να ασκείται και να αναπτύσσεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οι πτυχές που αφορούν ε, τους ανθρώπους, την ανάπτυξη. Επομένω, αυτά τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούσαν την Μπίργκετ. Και σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει το λόγο κάποιος ε, βουλευτής, έχει κάποια ερώτηση, κάποιος να υποβάλει. Όχι, σημαίνει μέρα χωρίς ερωτήσεις. Θέλει όμως το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Λούτσου ή άλλος της. Yes, uh, good um, Καλησπέρα. Εγώ ασχολούμαι στο DigiHome Home με τις συμφωνίες επανεισδοχής. Συμφωνώ με τα ευρήματα ε, σε ό,τι αφορά την επανεισδοχή. Εμείς προσπαθούμε Βάζομαι στις συμφωνίες επανεισδοχής την ε, κούσια επιστροφή. Είναι ένας ε, τρόπος που τον ε, προωθούμε για την επιστροφή οι συμφωνίες επανεισδοχής σημειώνεται ότι ε, παρέχουν καλή νομική βάση, αλλά οι πρακτικές λεπτομέρειες πρέπει να βελτιωθούν. Είχαμε παρόμοια ευρήματα στην αξιολόγηση των επανεισδοχών που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 2011. Επίσης θέλουμε να παρακολουθήσουμε την ε, κογούσια επιστροφή ε, με βάση τις χώρες Ουκρανία και Πακιστάν για να δούμε τι γίνεται μετά την επιστροφή. Το πρόγραμμα θα αρχίσει του χρόνου. Τέλος, πολύ σημαντικό, θέματα ε, ανάπτυξη τίθενται και επίσης οι μεταναστευτικές ροές με τρίτες, προς τρίτες χώρες, από τρίτες χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε Ενάπτυξη, παράδομη, νόμιμη μετανάστευση ε, είναι βασική πυλώνη της πολιτικής μας. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κασπάρεκ, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, εντάξει. Ε, ευχαριστώ λοιπόν. Σας πενθυμίζω ότι το σχέδιο της γνωμοδότησης θα ψηφιστεί στις 18 Δεκεμβρίου. Θέλει κάποιος να λάβει το λόγο για τα διάφορα. Κανείς. Ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης, δηλαδή καθορισμό της ημερομηνίας της επόμενης μας συνεδρίασης. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα γίνει στις Βρυξέλλες 18 Δεκεμβρίου από τις 9 στις 12.30 και από τις 3 ως 18.30. Αν θέλει ο Θεός βέβαια. Σας ευχαριστώ όλους και κλείνω τη συνεδρίαση της ε, σημερινής ημέρας. Αλλά ακολουθεί συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών για, την, ε, για τους δύο τριγωνικούς διαλόγους που είναι ένα εξελίξη για τον, ε, το εθελοντικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και συνεργασίας και εδώ μπορούν να είναι παρόντες μόνο οι βουλευτές της Επιτροπής μας, οι βοηθοί τους, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων και τα μέλη της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τρία λεπτά για να αποχωρήσουν ησύχως και σιωπηλώς τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονται στην αίθουσα. και σας παρακαλώ συνεχίστε τις συζητήσεις σας έξω για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ.